Σα everybody. Um, Σας καλωσορίζω και παρακαλώ να προσπαθήσετε να καθίσετε διότι έχουμε μεγάλο φόρτο εργασίας, πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας όπως πάντοτε γιατί είναι αυτή η προσπάθειά μας και νομίζω ότι δεν χρειάζονται εισαγωγές. Έτσι θα κερδίσουμε 5 λεπτά από τα 10 που χάσαμε. Εδώ έχουμε δημόσια κρόαση για τα παράγωγα και θα γίνουν παρουσιάσεις από επόπτες. και εκπροσώπους μεγάλων επιχειρήσεων και τις παρεμβάσεις αυτές θα τις ακούσουμε πρώτα και μετά θα γίνει γύρος ερωταπαντήσεων. Ο πρώτος μας ομιλητής, ο κύριος Ζούε, πρέπει μάλιστα να φύγει. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, θα προσπαθήσετε να κάνετε πρώτα ερωτήσεις προς εκείνον για να μπορέσει να φύγει έχοντας απαντήσει. Και θα καταλήξει ο εισηγητής μας για τα παράγωγα. Παρακαλώ λοιπόν τους ομιλητές και τις ομιλήτριες να σεβαστούν το χρόνο τους γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε χρόνο για ερωτήσεις και μπορεί να θυμώσουν οι βουλευτές. Και επίσης να μην μιλάτε πολύ γρήγορα διότι οι ερμηνευτές και οι ερμηνεύτριες θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες και θα χρειαστούμε και εμείς να σας διακόπτουμε για να λέμε πιο αργά, πιο αργά. Ο κύριος Ζαν Πιέρ Ζουέ που είναι πρόεδρος της Επιτροπής του Κέσαρος. Έχετε το λόγο κύριε Ζουέ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα περάσω κατευθείαν στην ουσία του θεματός και για να τα κάνω καλύτερα θα τα πω στα γαλλικά για να προσπαθήσω να πάω όσο μπορώ πιο γρήγορα. <clears throat> Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι κοινοβουλευτικοί, έρχομαι από το Λονδίνο και εκεί το σημερινό θέμα που συζητήθηκε ήταν ακριβώς αυτό το οποίο είχε αναφερθεί το Σεπτέμβριο το προηγούμενο στο Pittsburgh στις συνεδρίες των G20 το θέμα της τυποποίησης, της καταγραφής και του συμψηφισμού των παραγόγων εξοχρηματιστριακού χαρακτήρα. Σήμερα συνεδριάσουμε με στόχο να τηρήσουμε τα συμπεφωνημένα και είμαι πεπισμένος ότι θα μπορούσαμε πολύ γρήγορα να περάσουμε από τις αρχές στην πρακτική τους εφαρμογή. <clears throat> Ελπίζω λοιπόν ότι οι εργασίες σας, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο και την Κομισιόν, θα απολύξουν ταχαίως με συνεργατικό τρόπο, ώστε τα ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία θα καθορίσουμε να εμπνεύσουν αύριο και τους εταίρους μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που συναντώ και τον κύριο Λάγκεν, γιατί ήταν θαυμάσια η έκθεση την οποία έχει εκπονήσει και χάρη στην έκθεση του κύριου Λάγκεν έχουν εντοπιστεί, έχουν ε, ταυτοποιηθεί οι κύριες παράμετροι και οι χώροι όπου πρέπει να υπάρξει περαιτέρω εργασία. Χάρη στον κύριο Λάγκεν, το πιο δύσκολο κομμάτι της εργασίας έχει περατωθεί και οι ρυθμιστές των αγορών επίσης έχουν εργαστεί στα πλαίσια της ομάδος των ευρωπαϊκών ρυθμιστών των ε, αγορών αξιογράφων. Τι θέλουμε να πετύχουμε. Είναι κάτι το πολύ απλό. Θέλουμε σε περίπτωση πυρκαγιάς, δηλαδή σε περίπτωση που ε, πτωχεύει κάποιος συστημικός εταίρος, θέλουμε να έχουμε κάποιες θύρες πυρασφάλειας. Με άλλα λόγια, θέλουμε να μην επηρεαστούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ χρηματοοικονομικών εταίρων να οδηγήσουν σε διάδοση της κρίσης και να θέσουν σε κίνδυνο το σύνολο. Δεύτερον, δεδομένου ότι η διαφάνεια ευνοεί την καλή λειτουργία και την ολοκλήρωση των αγορών, θέλουμε επίσης να πετύχουμε κάτι το οποίο δεν είχε γίνει γεγονός μέχρι τώρα, να γνωρίσουμε ποιος αγοράζει τι, από ποιον και με τι τίμημα σε αγορές οι οποίες μέχρι τώρα ήταν απόλυτα διαφανείς. <clears throat> με ποιο τρόπο μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό. Νομίζω μέσω του τριπτύχου το οποίο προανέφερα, που είναι απαραίτητο για την ρύθμιση μετά από την χρηματοοικονομική κρίση, τυποποίηση, συμψηφισμό και καταγραφή σε Μητρώα. Καταρχήν το θέμα της τυποποίησης. Κάτι το οποίο είναι τυποποιημένο μπορεί να είναι εύκολα αντικείμενο συμψηφισμού. Βλέπουμε λοιπόν γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε κάτι τέτοιο, να έχουμε ένα κοινό πρότυπο, να έχουμε κοινά πρότυπα τα οποία επιτρέπουν να γίνεται με πιο αποτελεσματικό τρόπο ο συμψηφισμός. <clears throat> Ξέρουμε ότι δεν είναι τυποποιήσιμα όλα τα παράγωγα. Αυτό όμω δεν πρέπει να είναι λόγο για να μην προσπαθήσουμε να έχουμε φιλόδοξου στόχου σε ό,τι αφορά την τυποποίηση. Το θέμα του συμψηφισμού στη συνέχεια. Οι οργανισμοί συμψηφισμού είναι πράγματι θύρε πυρασφάλεια μέσα στο παράδειγμά μα. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω πόσο χρήσιμη είναι αυτή η φόρηση. Θέλω να τονίσω ότι αύριο θα είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος στο οικοδόμημα αυτό διαχείρισης του κινδύνου και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρουμε πρόσθετες προφυλάξεις για να είναι ισχυροί οι φορείς συμψηφισμού. Γι' αυτό το λόγο η ΣΕΖΑΡ, η Επιτροπή των Ευρωπαίων Ρυθμιστών των Χρηματαγορών, προτείνει φιλόδοξα πρότυπα για αυτούς τους φορείς συμψηφισμού. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να υπόκειται σε μια ρύθμιση ανάλογη αυτή των πιστοτικών φορέων. Μου φαίνεται σημαντικό αυτό, αλλά είναι η προσωπική μου άποψη και όχι η άποψη τη ΣΕΖΟ. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι απαραίτητο ένα φορέα συμψηφισμού να βρίσκεται στην, ε, στην χώρα όπου κυκλοφορεί το αντίστοιχο νόμισμα, ώστε να μπορεί να έχει γραμμή ρευστότητα από την κεντρική τράπεζα τη περιοχή με την οποία συνδέεται και που είναι ο δανειστή του φορέα αυτού, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Πρέπει επίσης να, να προσαρμόσουμε τις, επι... τις απαιτήσεις μας σε προληπτικό επίπεδο έναντι των τραπεζών, είτε συμψηφίζουν δεν συμψηφίζουν τις ε, συναλλαγές τους, να υπάρχει <clears throat> κάποιο... πρέπει να υπάρχει κάποιο πριμ στην περίπτωση του συμψηφισμού. Και αυτό προτείνει η Επιτροπή της Βασιλείας. Είπα ότι δεν μπορούν να τα να τύχουν τυποποίησης και Ω εκ τούτου δεν μπορεί να υπάρχει συμψηφισμό όλων των παραγόγων. Εξάλλου αυτό δεν είναι επιθυμητό γιατί υπάρχουν προϊόντα τόσο εξωτικού χαρακτήρα ώστε δεν υπάρχει να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου από τους φορείς συμψηφισμού. Τρίτο στοιχείο, η καταγραφή. <clears throat> δεν είναι φυσιολογικό και η κρίση για το κρατικό χρέος της Ελλάδος το κατέριξε ότι δεν είναι φυσιολογικό ένας ρυθμιστής να μπορεί με τρόπο άμεσο και χωρίς προβλήματα να γνωρίζει ποιες είναι οι συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην αγορά των παραγόγων. Τίθεται και ένα θέμα ευρωπαϊκής κυριαρχίας αλλά και ένα θέμα αποτελεσματικότητα στην εποπτεία των αγορών. Γι' αυτό η ΣΕΖΑΡ μελέτησε τη δημιουργία των λεγόμενων trade repositories, των μητρών συναλλαγών για τα παράγωγα που μας επιτρέπουν να έχουμε μια ενοποιημένη εικόνα των δεσμεύσεων και των ανοιγμάτων όλων των ε, παικτών της αγοράς για τα διάφορα προϊόντα. Ένα τέτοιο εργαλείο θα μπορέσει να βελτιώσει τη μακροπροληπτική ε, ε, εποπτεία των εξωχρηματιστριακών αγορών παραγωγών. Μπορεί να φανταστεί κανείς ότι αυτοί οι φορείς καταγραφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για στόχους μικροπροληπτικής εποπτείας για να μπορέσουν να διακριβώσουν και καταχρήσεις αγοράς. Και εγώ υποστήριζω μια τέτοια προσέγγιση. Θα μπορούσαμε να παραμείνουμε μονάχα στι ε, διατάξει τη οδηγία ΜΥΦ σε ό,τι αφορά τι εξωχρηματιστηριακέ αγορέ παραγωγών, σε ό,τι αφορά τι ε, εκθέσει προ το ρυθμιστή. Αλλά αυτό ο μηχανισμό είναι πάρα πολύ πολύπλοκο και επαχθή, γιατί αν έχουμε 27 ρυθμιστέ, είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε τη διασταύρωση των συλλεχθέντων πληροφοριών. Συλλεχθισών, μάλλον. Είναι καλύτερα να έχουμε ένα κεντρικό σύστημα συλλογή πληροφοριών μέσω των μητρώων συναλλαγών κάτω από ορισμένε συνθήκε, τα μητρώα αυτά θα μπορούσαν να δίνουν πληροφορίες και στους εμπλεκόμενους, στου συμμετέχοντες στις αγορές και όχι μονάχα στις ρυθμιστικέ αρχές σε σχέση με τις συνθήκες κατά τι οποίε έχουν γίνει ορισμένες συναλλαγέ. Αυτό είναι η λεγόμενη διαφάνεια μετά από την συναλλαγή. Σε ό,τι αφορά την τοποθεσία που θα πρέπει να είναι αυτή οι φορεί ε, καταγραφή και τον αριθμό του, υπάρχουν δύο απόψεις, δύο σχολές αν θέλετε. Θα έχουμε ένα ενιαίο μητρό συναλλαγών σε, ευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να έχουμε μια σαφέστερη και συνολικότερη εικόνα για τις συναλλαγές παραγόγων. Και δεύτερον, η δεύτερη άποψη λέει ότι πρέπει να είναι ένα τέτοιο μητρό συναλλαγής σε κάθε περιφέρεια που υπόκειται σε ενιαία ρύθμιση και επομένως θα έχει την εγγύηση μέσα σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση και περιοχή της διαφάνειας. Και οι δύο λογικές μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Εάν θέλουμε να είμαστε εξαντλητικοί στα θέματα αυτά, η φιλοδοξία μας θα πρέπει να είναι να υπάρχει ένα παγκόσμιο μήτρο συναλλαγών με την πρόσβαση φυσικά ότι ο Ευρωπαίος ρυθμιστής θα έχει πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα. Αν τώρα αυτό δεν μπορέσει να γίνει πραγματικότητα, θα πρέπει να έχουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ευρωπαϊκό χώρο, το δικό μας Μήτρο Συναλλαγών μέσα στον χώρο ενεργής, ε, ενεργών ε, συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα μπορούσαμε να δεχτούμε όλα τα, όλες οι συναλλαγές που γίνονται από ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς το φορείς να ελέγχονται και να είναι προσβάσιμες σε ένα εξωτερικό φορέα και εσείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είσαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο θέμα αυτό, πιστεύουμε σε αυτήν την περίπτωση ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να πριτανεύσει στα θέματα αυτά. Επομένως, τυποποίηση, συμψηφισμός και εγγραφή σε Μητρώα, αυτό είναι το πρόγραμμα εργασίας μας. Η ΣΕΖΑΡ ακολουθεί σε αυτά τα πλαίσια το φύλλο πορείας των G20 και ο στόχος μας είναι να περάσουμε όσο το δυνατόν την ε, εμπορία εξωχρηματιστηριακών παραγόγων σε οργανωμένες αγορές. Και πιστεύω θα ήταν ενδιαφέρον να προσθέσουμε σε αυτή την προβληματική το στοιχείο της ρύθμισης μετά από την χρηματοοικονομική κρίση. Κλείνον, θα ήθελα να σας δώσω την προσωπική μου άποψη για δύο θέματα για τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Λάγκεν καθώς και άλλοι κοινοβουλευτικοί έχουν να εκφέρουν γνώμη αλλά που δεν έχουν ακόμα ε, εξεταστεί σε βάθος από την Επιτροπή μας, την Επιτροπή των Ευρωπαίων Ρυθμιστών Αγορών Κινητών Αξιών. Καταρχήν ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκή, του Ευρωπαϊκής Αρχής Εποπτείας για τις κινητές αξίες και τις αγορές πιστεύω ότι θα πρέπει καταρχήν να έχει ένα πανευρωπαϊκό χαρακτήρα και να λειτουργεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να έχει και σχέσεις με τους εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι χρήσιμο λοιπόν σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Αρχή για τις Τράπεζες να είναι ο φορέας ο οποίος θα δίνει την έγκριση στους φορείς συμψηφισμού σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τους και να έχει και το δικαίωμα να παρακολουθεί τη λειτουργία τους. Δεν πιστεύω όμως ότι μπορεί να εφαρμόσει μια καθημερινή εποπτεία για την καθημερινή εποπτεία αυτών των φορέων συμψηφισμού πιστεύω θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει η επαφή και η διατηρία τους με τους εθνικούς επόπτες. Έχετε ξεπεράσει κατά ένα, χρόνο την, κατά ένα λεπτό το χρόνο παρέμβασή σας κύριε Ζουέ. Μπορείτε να περατώσετε. Τελευταία παρατήρηση μου φαίνεται σημαντικό η ΕΣΜΑ, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας, να μπορέσει να ελέγχει το σύνολο των χρηματοπιστωτικών φορέων, τράπεζες, ασφάλειες, χρηματαγορές και όλα αυτά και ιδίω δίνοντας την απαραίτητη προσοχή σε φορείς οι οποίοι δεν είναι καθαρά χρηματοοικονομικοί όταν υπάρχει μια ανάγκη εξαίρεσης. Τονίζω λοιπόν ότι εν ώψη της ανάγκης μητρών συναλλαγών και φορέων συμψηφισμού θα πρέπει να ξαναδούμε την οδηγία για τις αγορές ώστε οι ρυθμιστές να γνωρίζουν ποια είναι τα προβλήματα για αδικήματα λόγω χρήσης εσωτερικών πληροφοριών. Αυτά ήθελα να πω κυρία Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Έχει διανεμηθεί η ομιλία στις ε, πρωτότυπες γλώσσες, έχουν διανεμηθεί οι ομιλίες. Αν θέλετε να δείτε κάτι ξανά Και αν δείτε κάτι που ίσως ε, παρελήφθη από τον ε, ομιλητή για τον διάκοψα μπορείτε να δείτε το γαλλικό κείμενο. Εκ, πα, ο Ενρή Πόλσον παρέχει υποδομές στη Nasdaq OMX ε, παροχή παραγόγων. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου και κύριε Λάγκεν, ευχαριστώ πολύ να μιλήσω εκ μέρους των συμψηφιστικών φορέων και των χρηματιστηρίων. Είμαι ο Χένι Πόλσον, είμαι στην Nasdaq Comax, ασχολούμαι με τα παράγωγα. Η Nasdaq Comax είναι παγκόσμιος φορέας στα χρηματιστήρια και στους οίκους συμψηφισμού. Ε, λειτουργούμε σε αγορές όλο τον κόσμο και παρέχουμε και τεχνολογία στην αγορά σε πάνω από 70 αγορές, 50 χώρες. Πέρασα όλη μου την καριέρα στα παράγωγα χρηματιστήρια και σε οίκους συμψηφισμού. Τα παράγωγα είναι ένα φανταστικό μέσο, φανταστικά μέσα. Πάρα πολύ σημαντικά για εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, για μια σύγχρονη οικονομία. Όμως, και λυπούμε που υπάρχει ένα αλλά, ήρθε η ώρα να εστιαστούμε περισσότερο στη διαχείριση του κινδύνου και στην ρύθμιση και στον έλεγχο. Το 2008 η οικονομική αυτή κρίση Μα έδειξε με οδυνηρό τρόπο ότι τα παράγωγα αυτά, τα έξω χρηματιστηριακά, μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο στην οικονομία, εάν δεν τα χειριστούμε σωστά, επαρκώς. Οι συμμετέχοντες στην αγορά, οι τράπεζες, χρηματιστήρια, και συμψηφισμού και άλλοι φορεί μαζί με τους πολιτικούς και τις ρυθμιστικέ αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία και σημαντικότατα μέτρα για τη μείωση των κινδύνων στον τομέα των παραγόγων. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθώ στα συμπεράσματα που θα συναγάγουμε. Λοιπόν, και μπορώ να παραθέσω εδώ τι υπόθηκε. Όλα τα τυποποιημένα έξω χρηματιστηριακά παράγωγα θα πρέπει να είναι αντικείμενο συναλλαγέ σε ηλεκτρονικέ πλατφόρμε ή σε ε, χρηματιστήρια όπου ενδείκνεται. Και θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2012 το αργότερο να έχουν ε, καθαριστεί. Οι συμβάσεις θα πρέπει να αναφερθούν στα, στα μητρώα δεν θα πρέπει τα κεντρικά κατοχυρωμένα τέτοια συμβόλαια να υπόκεινται σε απαιτήσει υψηλότερε κεφαλουχικέ. Είναι πολύ σημαντική δήλωση αυτή που έγινε και είναι σημαντικό να εφαρμοστεί γρήγορα αυτή η αρχή από τους ε, G20. Θα είναι σημαντικό βήμα ε, για να αναπτύξουμε σταθερές χρηματοπιστωτικές αγορές και για να μπορέσει να ανακάμψει η ευρωπαϊκή οικονομία. Τα χρηματιστήρια και τα CCPs δημιουργήθηκαν εξυπηρετούν το στόχο μια σταθερή οικονομική χρηματοπροστατική αγορά. Ήταν πρόβαλαν αντίσταση, άντεξαν στην κρίση. Καθ' όλη τη διάρκεια τη κρίση τα χρηματιστήρια και άλλοι φορεί έδιναν πρόσβαση στου επενδυτέ σε διαφανεί και εύρυθμα λειτουργούσε αγορέ, παρήχαν εμπιστοσύνη και σταθερότητα σε ένα δοκιμαζόμενο οικονομικό σύστημα. Τα ωφέλη του, του κεντρικού κεντρικής εκαθάρισης οδηγούς, ε, οδηγεί σε καλύτερο έλεγχο τη αγορά ή ή Η οίκηση ψηφισμού ε, μπορεί και να πολλά και να πουλεί και να αγοράζει. Και έτσι ο συμψηφισμός σε κεντρικό επίπεδο επιτρέπει την σωστή συμμετοχή όλων των συμμετοχόντων και υπάρχει και η σωστή παροχή εγγυήσεων όσον αφορά τι διάφορε τοποθετήσει. Όσον αφορά τη δομή της αγοράς, αυτός ο οίκος συμψηφισμού σε κεντρικό επίπεδο είναι σε καλύτερη θέση οποιοδήποτε άλλο για να αξιολογήσει τον κινδύνο που απορρέει από τα παράγωγα. Αυτά τα κεντρικοί φορείς συμψηφισμού έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για αυτό τον σκοπό και θα ήθελα να τονίσω τρεις πολύ σημαντικές ε, πτυχές που καθιστούν τόσο σημαντικό σημαντικούς αυτούς τους κεντρικούς οίκους συμψηφισμού και είναι πολύ καλά δομημένοι. Γιατί το λέω αυτό. Πρώτα απ' όλα αυτοί και συμψηφισμού θέτουν ένα πλαίσιο πειθαρχημένο για τη διαχείριση του κινδύνου στην αγορά. Είναι μέσα στα γονίδια των οίκων συμψηφισμού αυτό. Πάντα να σκέφτονται τον κίνδυνο και το, τη διαχείριση του κινδύνου. Πάντα πρέπει να υπάρχουν εγγυήσει. Πάντα χρειάζεται ισότιμη αντιμετώπιση. Ποτέ να μην υπάρχουν εξαιρέσει για μεγάλου σημαντικού πελάτε έναντι μικρών πελατών, γειτόνων κλπ. Πάντα ίση αντιμετώπιση όλων. Πάντα να προσπαθούμε να αποκλείσουμε τις χρεοκοπίες. Θα πρέπει να δρουν μάλλον άμεσα αποφασιστικά η οίκηση ψηφισμού. Ακόμα και όταν υπάρχει υπόνοια κάποιες ε, πιθανότητες να μην πληρωθούν τα χρέη. Και αυτό είναι ο μεγάλος, η μεγάλη συμβολή των κεντρικών οίκων ψηφισμού. Ένα πλαίσιο ε, το οποίο είναι συγκεκριμένο το κεντρικό οικό ψηφισμού επιτρέπει ε, κάλυψη κάπως των κινδύνων. Να υπάρχει αντιστοιχεία συναλλαγών με τους συναλλασσομένους. Τα συμψηφίζει ο ψηφισμού όλα αυτά, τις συναλλαγές, μια γενική συναλλαγή με έναν ομόλογο. Τρίτο μοναδικό χαρακτηριστικό αυτών των κεντρικών οίκων συμψηφισμού ποτέ ποτέ δεν τοποθετούνται. Ποτέ δεν αναλαμβάνουν κίνδυνο τη αγορά. Αν υπάρχει κάποια θέτηση θέση υποχρέωση όπου υποχρεώθηκε κεντρικό 20 ψηφισμού να κινηθεί θα πρέπει να δράσει αμέσως για να κλείσει αυτή ε, ο φορέας που πραγματοποιεί αυτή την κίνηση. Αυτά τα χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα του κεντρικού ήχου συμψηφισμού ε, Κάνω αυτό το φορέα ιδανικό για διαχείριση του κινδύνου και είναι ισχυρότερο φορέα σε οποιαδήποτε άλλη διαθέτηση όπω είναι συμψηφισμό σε διμερέ επίπεδο. Όλων τούτων λεχθέντων και επενώντα του οίκου συμψηφισμού για του οποίου εργάστηκα επί μακρόν, αναγνωρίζουμε ότι κεντρικό οίκο συμψηφισμού ε, δεν είναι η ιδεώδη λύση για όλα τα προϊόντα. Υπάρχουν κάποια παράγωγα ε, που είναι πάρα πολύ περίπλοκα, πολύ υψηλού κινδύνου ή χρησιμοποιούνται σπάνια. Και αυτά τα προϊόντα ε, δεν πρέπει να ρυθμίζονται μέσω του κεντρικού οίκου συμψηφισμού. Ο κεντρικός οίκος συμψηφισμού μπορεί να επιφέρει μεγάλη συμβολή σε μεγάλο κομμάτι της αγοράς, δεν μπορεί να λύσει τα πάντα όμως, όλα τα προβλήματα της αγοράς. Όσο περισσότερα παράγωγα επεξεργάζεται αυτό ο κεντρικό φορέα ψηφισμού, θα πρέπει αυτοί οι φορεί να ρυθμίζονται με καλύτερο τρόπο όσο αυξάνονται οι υποθέσει που χειρίζονται. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο χρειάζεται ρύθμιση των κεντρικών οίκων συμψηφισμού. Θα πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό τμήμα τη νέα νομοθεσία. Αυτό θα δημιουργήσει και ισότιμε συνθήκε στην Ευρώπη για του οίκου συμψηφισμού. Και σαν Nasdaq Comex καλωσορίζουμε αυτό το γεγονό και σε επίπεδο ρυθμιστικό και σε επίπεδο εποπτείας των οίκων συμψηφισμού. Ισότιμες συνθήκες να επικρατούν στην Ευρώπη για όλους. Θα ήθελα να τονίσω μόνο κάτι, ένα πράγμα από τα πολλά που θα πρέπει να ρυθμιστούν για τους κεντρικούς οίκους συμψηφισμού. Πιστεύω ότι η ανεξαρτησία αυτού του φορέα είναι πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, ούτως ώστε να εξασφαλίζουμε αποφυγή συγκρούσεων όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων και ότι ο κεντρικό φορέα συμψηφισμού θα μπορεί να κινείται αυτόνομα στον τομέα της διαχείρισης των κινδύνων. Επίση, τα χρηματιστήρια μπορούν να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο, αυξάνοντα τη σταθερότητα της αγοράς. Προφανώ η διαφάνεια της τιμολόγησης μέσω συναλλαγών στα χρηματιστήρια ωφελεί γενικότερα το, οικονομικό, το χρηματοδοτικό σύστημα, απαιτώντα και κάποια παράγωγα εξοχρηματιστηριακά να περνούν από το χρηματιστήριο, τότε οι συναλλαγές θα γίνονται με τον πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο, με πλήρη διαφάνεια για όλους τους χρήστες. Πέραν αυτού, οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο δίνουν ουδέτερη και ανοιχτή πρόσβαση στις αγορές, κρισίμου σημασία σε αυτό και κυρίως σε περίοδο αναταραχής, όπου ο κόσμος θέλει ανοιχτές αγορές προσβάσιμες ε, για τους περισσότερους στο μέγιστο βαθμό μάλλον προσβάσιμος. And now a short note on uh, corporate... Και τώρα για τους τελικούς χρήστες των επιχειρήσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή και χρειάζονται κάποια συγκεκριμένη ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Έχουν ειδικέ ανάγκες αυτές οι επιχειρήσεις όχι όλοι οι τελικοί χρήστες, όλες οι εταιρείε θεωρούνται συστημικός κίνδυνος. Πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. Όμως, το θέμα του συστημικού κινδύνου δεν θα πρέπει να κρίνεται μόνο βάσει πώ κάποιο με τυπικό τρόπο χρησιμοποιεί τα παράγωγα, όχι με το πώ χρησιμοποιεί συνήθως τα παράγωγα. Υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι χρήση των παραγόγων και ίσως στην πράξη να είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθορίσει και να παρακολουθεί αυτή τη χρήση στην πραγματικότητα, στην καθημερινή ζωή. Ο καλύτερος τρόπος να προσμετρήσει κανείς ενδεχόμενο συστημικό κίνδυνο είναι μέσω μεγέθους. Πολύ μεγάλες σημαντικές θέσεις μπορούν να δημιουργήσουν συστημικούς κινδύνους ανεξάρτητα από τη φύση της επιχείρησης. Πιστεύουμε συνεπώς ότι πάνω από ένα επίπεδο εμπλοκής η κεντρική οι οίκοι συμψηφισμού θα πρέπει να ασχολούνται και με, τους, ε, με τις επιχειρήσεις που είναι τελικοί χρήστες των προϊόντων αυτών. Και επειδή τελειώνει η ώρα μου, ο χρόνος μου, ένα σύντομο συμπέρασμα, κάποια συμπεράσματα μάλλον, τα παράγωγα, τα εξοχρηματιστιακά ήταν στο επίκεντρο ε, της κρίσεως. Πρέπει να λάβουμε τα αναγκαία σημαντικά μέτρα για να μειώσουμε τους κινδύνους στον τομέα των παραγώγων των εξοχρηματιστηριακών θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι κανόνε και οι ρυθμίσει να δώσουν καλύτερα κίνητρα στην αγορά, να επιλέγουν ασφαλέστερου τρόπου εμπορία και συμψηφισμού ή και συμψηφισμού τα χρηματιστήρια και οι φορείς κατάθεσης και θα πρέπει να ε, αυξήσουν την ασφάλεια ε, του τομέα και να βελτιώσουν την, ε, το συνέστημα ασφαλείας στις χρηματιστηριακές αγορές στο μέλλον. Η διαχείριση του κινδύνου είναι σαν να προσπαθεί κανείς να πιάσει μια μαύρη γάτα σε ένα δυσκοτεινό δωμάτιο. Και η αυξημένη χρήση των οίκων συμψηφισμού δεν θα βγάλουν τη γάτα από το δωμάτιο. Θα ανάψουν το φως όμως. Και η γάτα, είναι πιο εύκολα να την πιαστεί η γάτα όταν αναμένω το φως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank ευχαριστώ. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να σεβαστεί κανείς το χρόνο του. ακούσαμε δύο ομιλητές και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Blythe Masters. Την κυρία. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Είμαι επικεφαλής των Global Commodities στην Jake Morgan, στην JP Morgan. Φυσικά είναι γνωστό ότι οι μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο και στη δημιουργία και στην αντιμετώπιση της κρίσης και πρέπει να πάρουμε τα μαθήματα που χρειαζόμαστε από αυτό. Τα παράγωγα βέβαια είναι αναπόσπαστο τμήμα της οικονομίας μας. Και έτσι θα τονίσω δύο θέματα που, ταύτισαν, που ταύτισε ο εισηγητής. Πρώτον, ότι δεν υπάρχουν σαφείς υποδομές συμψηφισμού και δεύτερον δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια, ιδίως για τους ρυθμιστές. Η κερδοσκοπία έχει αναφερθεί πολλές φορές και ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της είναι η δημιουργία μιας κεντρικής υπηρεσίας συμψηφισμού. Αυτό όμως θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη του δύο παράγοντες. Πρώτον, δεν μπορούν όλοι να συμψηφίσουν τη δραστηριότητά τους. Και ο υποχρεωτικός συμψηφισμός θα υποχρέωνε μερικές επιχειρήσεις ε, μέχρι και να κλείσουν λόγω του υψηλού κόστους. Δεύτερον, δεν μπορούν όλα τα παράγωγα να συμψηφιστούν, διότι για να υπάρξει σωστή διαχείριση μόνο όταν είναι αρκετά ρευστά τα παράγωγα μπορούν να συμπληφιστούν. Ναι, ναι, θα, θα τα λέω πιο αργά, πιο αργά. Λοιπόν. Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί τρέφουν το σύστημα και οι περισσότεροι χρήστες τους δεν ε, αντιμετωπίζουν ούτε δημιουργούν ιδιαίτερο συστημικό κίνδυνο. Ο κοινό μας στόχο μείωση του κινδύνου θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερα με μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ ε, θεσμών ή θεσμικών οργάνων που χρησιμοποιούν παράγωγα. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι το μεγαλύτερο τμήμα των παραγόγων στην αγορά θα γινόταν ελαστικό και πιο διαφανές και θα υπήρχε κάποια όχι υπερβολική τυποποίηση εφόσον υπάρχει βέβαια και το κίνητρο για την τυποποίηση αυτήν. Θα ήθελα να συζητήσω ορισμένες προτάσεις για την, τον συνδυασμό των διαφόρων μεθόδων που υπάρχουν ψηφισμού. Τα ομόλογα και άλλες μορφές χρηματοδότης και παραγόγων δεν είναι όλα όμοια μεταξύ τους στη λειτουργία τους. Τα παράγωγα εξορισμού δημιουργούν περισσότερους κινδύνους και άρα πρέπει να υπάρχει διαφορετική μέθοδος υπολογισμού και του συμψηφισμού τους. Έχουμε λοιπόν μεγάλες αμφιβολίες από το κατά πόσον μία υπηρεσία συμψηφισμού θα μπορούσε να εφαρμοστεί. However, while there is an understandable rationale for imposing higher η ρύθμιση, η αντιμετώπιση του κεφαλαίου είναι το κλειδί για όλα αυτά και πιστεύουμε ότι για να μειωθούν οι κίνδυνοι μέσω διμερού συμψηφισμού θα έπρεπε να δούμε ότι αυτό είναι συγκρίσιμο με τον κεντρικό συμψηφισμό αλλά είναι πιο δύσκολη η υπολογισμή απλώς. Στην έκθεση Χάρης που πρόκειται να συγγραφεί θα αναφέρονται όλα αυτά πιο λεπτομερώς. Πρέπει να δούμε και ποιες θα είναι οι διοικητικές επιτροπές των διαφόρων οίκων συμψηφισμού. Πρέπει εκείνοι που ασχολούνται με τη διαχείριση της αγοράς και των παραγόγων να παίζουν κάποιο ρόλο και στους οίκους συμψηφισμού. Έτσι κατά κάποιον τρόπο οι παράγοντες της αγοράς θα κάνουν αυτοδιαχείριση και αυτοσυμψηφισμό και θα μειώνονται έτσι εξορισμού οι κίνδυνοι. Τώρα για τη διαφάνεια. Υποστηρίζουμε ολόψυχα τις προσπάθειες περισσότερης διαφάνειας για να μειωθεί ο συστημικός κίνδυνος και να λειτουργήσει καλύτερα η αγορά με λιγότερους κινδύνους. Παρ' όλα αυτά η διαφάνεια δεν είναι παρά ένα μέσο και όχι ένας αυτοσκοπός. Και γι' αυτό πρέπει να στοχεύσουμε καλύτερα τις στόχους μας για τη διαφάνεια μεταξύ των οποίων είναι και η διατήρηση της ρευστότητας. για να διασφαλίσουμε μια σωστά λειτουργούσα αγορά με, καλό, με καλή διαχείριση του κινδύνου πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα και της ρευστότητας και της διαφάνειας. Υπάρχει όμως ένα σημείο μετά από το οποίο μπορεί όλα αυτά να καταλήξουν αρνητικά. Γι' αυτό δεν θα θέλαμε να υπάρξει μεταφορά όλων των συναλλαγών σε, αυτά τα, σε αυτούς τους κεντρικούς οίκους συμψηφισμού. Ξέρω ότι συζητιέται αυτή τη στιγμή το θέμα της κερδοσκοπίας ως τμήμα της κανονικής λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι δεν μπορούμε να εμποδίσουμε κάποιο βαθμό κερδοσκοπίας νομοθετικά. Η δυνατότητα συναλλαγών είναι το ίδιο σημαντική με την δυνατότητα που πρέπει να έχει η επιχείρηση να αυτοπροστατευτεί. οι αγορές υπάρχουν επειδή υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες και απόψεις. Μερικοί το λένε αυτό επένδυση, άλλοι κερδοσκοπία. Αλλά αν το τελικό αποτέλεσμα είναι να μειωθεί η ρευστότητα και ο τελικός χρήστης, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε πετύχει το στόχο μας. Α, δεύτερος στόχος είναι να μην αυξάνονται τα ελλείμματα στου προπολογισμού των κυβερνήσεων ή να μπορούν οι κυβερνήσεις να τα χρηματοδοτήσουν. Και πάλι, αν περιορίσουμε τη δυνατότητα των επενδυτών να επενδύσουν ελεύθερα, μπορεί να μειώσουμε έτσι την εμπιστοσύνη της αγοράς και τελικά να αυξήσουμε το κόστος για τον φορολογούμενο και τη φορολογούμενη. Τέλος, υποστηρίζουμε τις περισσότερες συστάσεις της εκθέσης Λάγκεν. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ και καταφέρατε να τελειώσετε με μόνο δύο λεπτά. <laughs> Με δύο, δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του χρόνου σας. Νομίζω ότι αξίζει να σας χειροκροτήσουμε. Και ερχόμαστε τώρα στον ε, ε, επικεφαλής της ε, Deutsche Bank, ο οποίος θα πρέπει να μιμηθεί την κυρία Μάστερς γυναίκε θα καταφέρουν καλύτερα, επισημαίνει πρόεδρο. Κυρία Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να μιλήσω ενώπιον σα για το σημαντικό θέμα των εξοχρηματιστιακών παραγόγων. Εγώ θα εστιάσω στις αγορές των εξωχρηματιστιακέ αγορές και στι αλλαγέ που χρειαζόμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε μια καλά ρυθμισμένη αγορά για τα προϊόντα αυτά ξεκινώ με το γενικό πλαίσιο. Οι εξωχρηματιστηριακές, εξωχρηματιστηριακά παράγωγα υπάρχουν εδώ και 25 τουλάχιστον χρόνια και είναι ένας από τους ε, πρότυπους τρόπους με τους οποίους οι εταιρείε στην Ευρώπη διαχειρίζονται κινδύνους. Κινδύνους για συνάλλαγμα, κινδύνους που έχουν να κάνουν με συνεργασία με πολυεθνικές εταιρείε, το κόστος που έχει να κάνει με πολλαπλούς δανειστές, η Επίση, τα ταμεία συντάξεων και οι ασφαλιστικέ εταιρείε πρέπει να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά. Δίνουν λοιπόν στι επιχειρήσει ένα αποτελεσματικό μηχανισμό μεταφορά του κινδύνου για να εξασφαλίσουν υγεία χρηματοοικονομικά πλαίσια. Μεταφέρουν λοιπόν από του τελικού χρήστε, οι οποίοι δεν θέλουν να τα αναλάβουν, σε τράπεζε και άλλου φορεί στην αγορά που είναι ειδικευμένοι στην ανάληψη κινδύνων. Στην Ευρώπη έχουμε αποτελεσματικέ και ανταγωνιστικέ αγορέ εξοχρηματιστικών προϊόντων και αυτό είναι προς όφελος των εταιριών μας και των πολιτών μας. Αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να πράξουμε ορισμένα πράγματα και η, ο κλάδος θεωρεί ότι είναι μεγάλο καθήκον του να συνεχίσει τις προσπάθειες αυτές μαζί με τους ρυθμιστές και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Θα σταθώ σε τρία θέματα που είναι ο συμψηφισμός, η διαφάνεια και οι συναλλαγέ. Ξεκινώ με, την, με το συμψηφισμό και την παροχή εγγύησεων. Οι οίκοι συμψηφισμού, οι οποίοι έχουν ισχυρό κεφάλαιο και έχουν ε, ισχυρέ διαδικασίε ενόψη των αθετήσεων είναι κάτι το οποίο μπορεί να μειώσει τη δυνατότητα τη συστημική να υπάρξει μια γενικότερη κρίση και κατάρρευση. Ένα από του στόχου των ρυθμιστών και των νομοθετών στην Ευρώπη και στι ΗΠΑ είναι να αυξηθεί το ποσοστό των συναλλαγών εξοχρηματιστιακών προϊόντων που την χάνουν κεντρικού συμψηφισμού. Αυτό είναι λογικό <clears throat> για συστημικά επικίνδυνου χρηματοπιστωτικού φορεί, αλλά αυτό δεν έχει μεγάλο νόημα για πολλού τελικού χρήστε όπου είναι πολύ μεγαλύτερα τα προβλήματα τη ε, πολυπλοκότητα ενό τέτοιου μηχανισμού. Οι μη χρηματιστηριακοί φορεί γενικά δεν χρησιμοποιούν εγγύησει όταν κάνουν ε, συναλλαγέ OTC και δεν χρειάζεται επομένω να χρησιμοποιούν χρήματα ή να αντιμετωπίζουν την πολυπλοκότητα αυτή τη διαδικασία. Και εάν δεν το πράξουν, δεν θα έχουν τη δυνατότητα αντισταθμιση κινδύνου και θα πρέπει να υπομειστεί τον κίνδυνο αυτό η πραγματική οικονομία. Ένα άλλο θέμα το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να το λάβετε υπόψη σα είναι το να εξασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία θα καλύψει μόνο τα σωστά προϊόντα. Ορισμένα προϊόντα εξοχρηματιστιακά δεν προσφέρονται για συμψηφισμό γιατί δεν υπάρχει το βάθο αγορά για να μπορέσει να εξασφαλίσει το κόστο τη δημιουργία ενό φορέα συμψηφισμού ή όπου υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι που είναι πιο σημαντικοί. Αυτό είναι, για παράδειγμα, είναι η, η ανταλλαγή συναλλαγμάτων όπου ο κίνδυνο του διακανονισμού είναι μεγαλύτερο από τον κίνδυνο αντισυμβαλωμένου. Πρέπει λοιπόν να λειτουργήσουν από κοινού οι φορεί συμψηφισμού, ώστε και οι ρυθμιστέ για να δούμε ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο να πετύχουμε αυτά τα πράγματα. Είναι επίση λογικό τα μέλη αυτών των οίκων συμψηφισμού να έχουν κάποια συμμετοχή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι φορεί αυτοί. Θα κάνω τώρα ένα τελευταίο σχόλιο για τα θέματα αυτά. Πρέπει να υπάρξει σωστή ρύθμιση για τους φορείς συμψηφίσμου. Είναι απαραίτητο να μην συμμετέχουν σε ένα αγώνα προς τα κάτω σε σχέση με τα πρότυπα και να έχουν χαμηλότερα ε, επίπεδα εγγύσεων για αυτό το σκοπό. Διαφάνεια τώρα. Το κύριο θέμα τη διαφάνεια είναι ότι οι αγορέ OTC υπήρξαν αδιαφανεί για του ρυθμιστέ για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Για να υπάρξει αποκάλυψη τιμών πριν από τι συναλλαγέ, υπάρχουν αρκετά στοιχεία τα μπορούμε να βοηθήσουν του συμμετέχοντες στην αγορά να καταλάβουν ποια είναι μια εύλογη τιμή για αυτά τα προϊόντα. Και ο κλάδο μα δουλεύει με του ρυθμιστέ σε παγκόσμιο επίπεδο για να μπορέσει να τεκμηριώσει αυτά τα στοιχεία. Πιστεύω λοιπόν ότι η αποκάλυψη τιμών είναι ένα πρόβλημα στις αγοράς μα. Οι συναλλαγέ όμω και η κατάσταση μετά τι συναλλαγέ είναι πιο πολύπλοκη. Εμεί υποστηρίζουμε απόλυτα την πλήρη πρόσβαση για του επόπτε και προσπαθούμε να το επιτύχουμε αυτό για όλες τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού. Ένα παράδειγμα είναι το αποθετήριο συναλλαγών στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο υπάρχει από το 2006. Έχουμε ένα αντίστοιχο μητρό για τα επιτόκια στη Στοχόλμη και υπάρχουν σχέδια για, το, για ένα αποθετήριο σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές μετοχών στο Λονδίνο. Όλα αυτά είναι στοιχεία μιας γενική ε, λύσης, αλλά αυτό που είναι σημαντικό να υπάρχει πλήρης πρόσβαση για τους ρυθμιστές και τους επόπτες και υπάρχει μια πρόοδος για τα θέματα αυτά. Η δημόσια αποκάλυψη όμως των συναλλαγών σε όλους είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποβεί σε βάρος της ρευστότητα. Επομένω η ευρωπαϊκή ρύθμιση που αναγνωρίζει με την ε, οδηγία MIFID αυτό το θέμα και συνεχίζει να το πράττει θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν δημιουργήσουμε το νομοθετικό πλαίσιο για, τις για τα εξοχρηματιστηριακά παράγωγα. Έρχομαι τώρα για το θέμα της εμπορίας και της προτυποποίησης. Χρησιμοποιείται πολύ η έννοια προτυποποίησης για, τις, ε, για τα παράγωγα τα εξοχρηματιστηριακά. Αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι να υπάρχει τυποποίηση στη διαδικασία και στο νομικό πλαίσιο που θα οδηγήσουν σε μια αποτελεσματική αγορά. Σε ορισμένε περιπτώσει το να έχουμε στάνταρ προϊόντα μπορεί να έχει νόημα. Παραδείγματο χάρη, ε, συμφωνίες μελλοντικής εκπλήρωσης σε χρηματιστήρια. Αλλά για ορισμένα παράγωγα δεν έχει νόημα να είναι τυποποιημένα. Θα πρέπει οι χρήστες να μπορούν να τροποποιήσουν και να προσαρμόσουν τα παράγωγα αυτά στις πραγματικές τους ανάγκες. Συνεχίζεται λοιπόν το έργο μας στις αγορές OTC και ο συμψηφισμός, η διαφάνεια και η τυποποίηση μπορεί να μας βοηθήσουν να έχουμε τις καλύτερες επιμέτρων λύσεις σε ένα αποτελεσματικό τρόπο. Εν κατακλείδη, θέλω να πω τα εξής. Όλοι συμφωνούν ότι χρειάζεται να υπάρξει μια αναθεώρηση των χρηματαγορών για να μην επανέλθουν οι κλειδονισμοί που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Οι αγορέ εξοχρηματιστηριακών προϊόντων θα πρέπει να τιμήμα αυτή τη διαδικασία. Αλλά έχω τρία κύρια συμπεράσματα τα οποία θέλω να τονίσω. Πρώτον, πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια αυτών των αγορών, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με ένα προσεκτικό τρόπο για να μην θίξουμε την ρευστότητα των αγορών. Δεύτερον, συμψηφισμό είναι αποτελεσματικό τρόπο να μειώσουμε το συστημικό κίνδυνο, αλλά αν υπάρχει μεγάλο άχθο για του τελικού χρήστε, αυτό δεν θα είχε νόημα γιατί οι τελικοί χρήστε δεν έχουν συστημικό κίνδυνο. Τρίτον, οι αγορέ ε, δεν μπορούν να καλύψουν όλα τα εργαλεία διαχείριση των ε, τελικών χρηστών και ο καλύτερο τρόπο να καλύψουν αυτού του κινδύνου πολλέ φορέ είναι εξωχρηματιστιακά παράγωγα. Πρέπει να συνεπάρχουν λοιπόν τα δύο είδη αγορά και σα ευχαριστω 33 λεπτά έχω ακόμα. Προφανώ. Έπρεπε να σα θέτω τι προκλήσει πιο συχνά. Προχωρούμε. Ας δούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι καλά. Με μεγάλους τελικούς χρήστες επιχειρήσεις. Το επόμενα 7,5 λεπτά, να δούμε αν θα τα καταφέρετε, να συνεχίσετε το καλό παράδειγμα, κάποιος το οποίο το όνομα δεν μπορώ να προφέρω. Είναι ο Χέκαν Φινκ, ε, διευθυντής του Market Rules για τη στρατηγική στα ενεργειακά προϊόντα. Ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσω για αυτό το θέμα. Το εμπόριο ενέργειας είναι πολύ σημαντικό θέμα. Οι μεγάλοι καταναλωτές και οι παραγωγοί θα μπορέσουν να αποφύγουν να πεθούν ε, σε πτυτικότητα και οι λιανοπολιτές θα μπορούν να προστατευθούν ε, έναντι της πτυτικότητας των τιμών απέναντι στους καταναλωτές. Οι αναπτυσσόμενες αγορές αερίου, αερίου και ηλεκτρισμού είναι αναπτυσσόμενες αγορές για την Ευρώπη ε, και ο ανταγωνισμός θα οδηγεί σε ανταγωνιστικές τιμές στον τελικό χρήστη. Οι αποφάσεις, οι πολιτικές όσον αφορά τα εξοχρηματιστικά παράγωγα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικέ ανάγκες αυτών που εμπορεύονται αυτά τα προϊόντα, που προσπαθούν να προστατεύσουν κάποια πράγματα. Θα πρέπει αυτό να συνάδει με την ανάγκη ε, την, τον, που έχουν οι οι αγορές ρευστής ενέργειας. Χρειάζεται τυποποίηση που θα βελτίουν ε, τον έλεγχο, το ρυθμιστικό. Ε, ο υποχρεωτικός συμψηφισμός και ο υποχρεωτικές συναλλαγές εντός χρηματιστηρίου αυτών των προϊόντων, αυτών των παραγόγων του τομέα μας προβληματίζει. Ε, συστημικά τα παράγωγα, τα εξωχρηματιστηριακά ίσως να προστατεύουν τους τελικούς χρήστες έναντι της ανάλογης χρήσης των προϊόντων. Εκ, αντίθετα το χρηματιστηριακό τομέα, αν μια εταιρεία που παρέχει ενέργεια έχει περιορισμένες ε, συνέπειες όσον αφορά τις τιμές. Το είδαμε πρόσφατα όταν είχαμε ε, χρεοκοπίες σημαντικών φορέων. Η ένωρων παραδείγματος χάρη είναι ένα παράδειγμα ε, του τομέα. Ο τελικός χρήστης προστατεύεται, αυτό είναι σημαντικό. Από τη ρύθμιση των ενεργειακών αγορών. Εξασφαλείται φυσική ασφάλεια και συνεχής εφοδιασμός ε, όταν υπάρχει πρόβλημα στην ενεργειακή αγορά. Δείτε τη διαφάνεια που παρουσιάζω εδώ, που ίσως να εξηγεί πώς ασχολούμαστε και αντιμετωπίζουμε διαχείριση του κινδύνου. Ο τομέας της ενέργειας ε, χρειάζεται μεγάλα κεφάλαια ε, και χρειάζονται επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ενέργειας και υπάρχει έκθεση και δημιουργείται κίνδυνος. Αυτό χρειάζεται πλαίσιο να περιορίσουμε ε, χρειαζόμαστε όρια όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων, την, ε, τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει η πίστοση και η ροή του κεφαλαίου. Χρειάζεται ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την αντιμετώπιση του κινδύνου. Αν εστιαστούμε σε έναν τομέα από όλου, παραδείγματο χάρη, ε, τα, θα γνωρίσουμε τον, τους άλλους δύο από το τρίγωνο. Έχουμε αυστηρέ πολιτικές για τις πιστώσεις και η πίστοση, όσον, όσον αφορά εκείνη την πίστοση, πρέπει να είναι σε αποδεκτό επίπεδο βελτιστοποιούμε το εμπόριο έξω ε, ε, χρηματιστηριακά, χρηματιστηριακά δημιουργούμε ένα σωστό κράμα. Παραδείγματο χάρη, μία μονάδα παραγωγής από άνθρακα ε, γίνεται, προστατεύομαστε τον κίνδυνο πουλώντας, πουλώντας το ηλεκτρικό ρεύμα αγοράζοντας άνθρακα. Οι συναλλαγές γίνονται είτε σε χρηματιστήρια είτε στην έξω χρηματιστηριακή αγορά ανάλογα με την αξιολόγηση του κινδύνου και επίσης είμαστε διαφανείς όσον αφορά την έκθεσή μας. Δημοσιεύουμε την ετήσια έκθεση ε, βάσει των ε, κινδύνων τιμολόγησης. Λοιπόν, στο 20 ψηφισμού πρέπει ε, να καταθέσουμε χρήματα. Όταν αλλάζει η τιμή της αγοράς, αλλάζει το, η τιμή, το χρήμα που πρέπει να διαθέσουμε για την προστασία από τον κίνδυνο. Εάν υποχρεωτικά περνάμε από 20 ψηφισμού, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα για τον τελικό χρήστη. Ο κίνδυνος για τις τιμές ή για την οικονομική ροή θα αυξηθεί αν υπάρχει υποχρεωτική διέλευση μέσω του 20 ψηφισμού, διότι δεν μπορούμε να πετύχουμε βελτιστοποίηση. Αν αποφασίσουμε να έχουμε σταθερό το κίνδυνο στο φάση τιμές, θα έχουμε μεγαλύτερο κίνδυνο για τη ροή του ε, ρευστού Άρα θα πρέπει να έχουμε στο αποθεματικό περισσότερο ρευστό και δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό για, τα, για επενδύσεις και για τα λειτουργικά έξοδα. Οι τιμές έχουν διαφορετικά αποτελέσματα και θα πρέπει να έχουμε στο απόθεμα ε, κάποια, κάποιο ρευστό για, αν υπάρξουν μεγάλες ανάγκες στην αγορά. Και αν θέλουμε να σταθεροποιήσουμε τον κίνδυνο για την ροή του ρευστού πρέπει να έχουμε λιγότερο αποθεματικό, αυξάνεται το επίπεδο του κινδύνου και έχουμε και λιγότερα χρήματα για επενδύσεις. Αν συγκρίνουμε αυτό με τα χρηματοστατικά ιδρύματα, βλέπουμε δύο βασικές διαφορές όσον αφορά τις συνέπειες των αντίκτυπων. Σαν τελικός χρήστης έχουμε μια φυσική θέση η οποία απορρέει από τις επενδύσεις μας. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που η τιμή του ηλεκτρικού αυξηθεί, ε, το, το απόθεμα θα αυξηθεί. Είναι διαφορετικό για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κανονικά είναι ουδέτερα. Και η δεύτερη διαφορά είναι ότι οι τράπεζες έχουν ευκολότερη πρόσβαση ε, στο ρευστό από ότι οι μη χρηματοπιστωτικέ εταιρείε. Για μα. θα δανείζαμε περισσότερα και θα άλλαζε το μητρό υπολογισμού και θα κάναμε καλύτερες ε, επενδύσεις. Σαν επιχείρηση ενεργειακή πρέπει να δούμε ποια είναι η εξέλιξη στην ενεργειακή αγορά. Οι αγορές σε πολλά μέρη της Ευρώπης δεν είναι ρευστέ ακόμα, δεν έχουν ρευστότητα. Και με υποχρεωτική διέλευση από συμψηφισμό αυξάνεται το άχθος όσον αφορά του εμπορευόμενους ενέργεια και θα δημιουργούνται φραγμοί για νέες επιχειρήσεις και αυτό είναι μια επώδυνη εξέλιξη. Τώρα, ε, δεν, έχουμε, δεν είμαστε σημαντικοί για το χρηματοδοτικό σύστημα, εμείς που εμπορευόμαστε αυτά τα προϊόντα, οι εμπορικές συναλλαγές ε, χρησιμοποιούνται για να μειώσουν τον κίνδυνο προσέγγιση μας. Οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο να δουν κατά πόσο δεν έχουμε κάποια θέση στην εξωχρηματιστηριακή αγορά, διότι αυτό θα συνεπάγεται ότι δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τη θέση μας. Το ίδιο ισχύει και για τις κεφαλουχικές απαιτήσει Εάν υπάρχουν αυτές οι απαιτήσει για μη ξεκάθαρες συναλλαγές να περνάμε από το 20 ψηφισμού, ε, η προσέγγιση δεν θα είναι ανάλογη. Όπως ήδη αναφέραμε στην αρχή, συμφωνούμε ότι η διαφάνεια πρέπει να βελτιωθεί. Θα θέλαμε να δούμε και εμείς τη γάτα και είναι σημαντικό οι ρυθμιστικές αρχές να ξέρουν ακριβώ τι συμβαίνει στην αγορά. Βλέποντας τις θέσεις από μια εταιρεία όπως είναι η δική μα, είναι σημαντικό να δούμε και ποια είναι τα στοιχεία του ενεργητικού, διότι χρησιμοποιούμε τα παράγωγα για να προστατεύσουμε την οικονομική μας θέση. Τώρα στα συμπεράσματα. Κατά την άποψή μα η διαχείριση του κινδύνου δεν θα πρέπει να βρει εμπόδια, θα πρέπει επιχειρήσει να ενθαρρυνθούν να κάνουν συναλλαγέ με διαχείριση του κινδύνου, είναι προ όφελο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη ασφάλεια εφοδιασμού, τιμέ για του τελικού καταναλωτέ και ευμάρεια και ασφάλεια για την Ευρώπη. Να εξασφαλίζουμε μάλλον μελλοντική ευμάρεια για την Ευρώπη. Υπάρχει ανάγκη για συμψηφισμό για συναλλαγές μεταξύ δύο χρηματοστατικών ιδρυμάτων και μόνο. Και θα θέλαμε τέλος να τονίσουμε ότι συνεχίζεται η δουλειά στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας για ένα καθεστώς για διαφάνεια και ρύθμιση της αγοράς του ενεργειακού τομέα. Και είναι μια αναλογική ρύθμιση που νομίζω θα ήταν επωφελής για τις αγορές. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλος ο Ρίτσαρντ Ρέιμπορν που είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συλλόγου ε, Ταμιών Επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Θα σας εξηγήσω καταρχήν γιατί ενδιαφερόμαστε για το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊ... Ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος ε, που αντιπροσωπεύω αντιπροσωπεύει επαγγελματικά σώματα και δεν είναι ομάδα πίεσης. Έχουν συμβεί μεγάλες αλλαγές, παραδείγματος χάρη πρώτα η ΣΕΠΑ και τώρα το θέμα του OTC. Εμείς ενδιαφερόμαστε για ένα απλό θέμα. Όπως φάνηκε από την αρχή, είδαμε ότι η εφαρμογή των προτάσεων θα ε, άδειαζε τα μία της Ευρώπης και αυτό θα μπορούσε να, κατα... να καταντήσει να αντιστρατεύεται το στόχο που είχαμε δηλώσει. είναι προφανώς πολύ σημαντικό να μιλήσουμε με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Εμείς είμαστε υπέρ των δεσμεύσεων που ανέλαβε το ΓΑΜΑ 20. Αυτά που ανέφερε ο Υπουργός ε, Γκάιτνερ πρόσφατα δείχνουν σαφώς πόσο καταστροφική ήταν η κρίση στη Wall Street. Όλοι θέλουμε να υπάρχουν ασφαλείς και βιώσιμες θέσεις εργασίας. Και το τονίζω αυτό γιατί θεωρώ ότι τα παράγωγα υποστηρίζουν την απασχόληση και την ανάπτυξη και ότι μειώνουν τον κίνδυνο, δεν τον δημιουργούν ούτε τον αυξάνουν. Πιστεύω ότι θα χάναμε ρευστότητα από τις προτάσεις ως έχουν. Και θα αφήναμε τις επιχειρήσεις πιο εκτεθειμένες στις κινήσεις, σαν ανεξέλεγκτες κινήσεις της αγοράς. Το σχέδιο έκθεση του κυρίου Λάγκεν αναφέρει πολλά σημαντικά προβλήματα, καθώς και οι τροπολογίες. Εγώ θεωρώ τέσσερα θέματα ως κύρια. Γιατί και πώς χρησιμοποιούνται τα παράγωγα τρίτον το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τέταρτον ποια αποτελέσματα έχουν όλα αυτά στην πραγματική οικονομία της Ευρώπης. Δεν εννοώ την κερδοσκοπία, ε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ποιος ακριβώς είναι ο κίνδυνος που περιέχουν τα παράγωγα. Σχετίζεται με τα επιτόκια και τις νομισματικές ισοτιμίες γιατί οι εταιρείε και εισάγουν και εξάγουν. Έχω εργαστεί και σε μεγάλες και σε μεσαία διαστάσεων επιχειρήσεις στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία και ξέρω ότι ένα διοικητικό συμβούλιο πάντοτε θέλει να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο. Και αυτό φαίνεται και από πολλά πολιτικά προγράμματα και δηλώσεις. Μερικοί λένε ότι το hedging είναι κερδοσκοπία. Η απάντησή μου είναι απλή. Το hedging, δηλαδή η μείωση του κινδύνου, δημιουργεί βεβαιότητες, ενώ αλλιώς θα υπήρχαν αβεβαιότητες στη θέση του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα κρατικό κατάστημα, πολυκατάστημα που όπου δουλεύουν 24.000 άνθρωποι. 25% του αποθέματός του εισάγεται σε δολάρια. Άρα είναι ουσιώδες να μειωθεί ο κίνδυνος εκεί. Έτσι, εκεί έρχονται τα παράγωγα. Ο τελικός χρήστης πρέπει να γνωρίζει, να έχει κάποια εγγύηση για το ποιο κίνδυνο εμπεριέχεται στη χρήση των, ε, από τη δραστηριότητά του. Οι εταιρείε χρησιμοποιούν τα παράγωγα και για να υπάρξει πιο αποτελεσματική διαχείριση πολλές αγγλικές εταιρείες χρησιμοποιούν τα παράγωγα για να εκμεταλλευτούν την ισοτιμία μεταξύ λίρας και δολαρίου. Θα ήθελα να τονίσω ότι εδώ δεν υπάρχει κανένα στοιχείο κερδοσκοπίας σε αυτήν τη χρήση των παραγόγων. Τρίτο θέμα. Οι χρήστες παραγόγων δημιουργούν συστημικό κίνδυνο. Νομίζω ότι αυτά είναι αποκοιήματα φαντασίας. Η πραγματική οικονομία δεν δημιουργεί μεγαλύτερο συστημικό κίνδυνο από τα παράγωγα και αυτό το έχω δει και στην πράξη. Έχουμε δει πώς μπορεί να αποτύχει μια τράπεζα μέσα σε ένα και μόνο Σαββατοκύριακο Τα γνωρίζετε τα ονόματα Lehman Brothers κλπ. Και τα ονόματα που αναφέρω δεν απέτυχαν λόγω συστημικού κινδύνου. Οι τράπεζες δεν αποτυγχάνουν επειδή εκτίθενται σε μεμονωμένες εταιρείες επιχειρήσεις. Και γι' αυτό θεωρώ ότι η κατηγορία ότι η χρήση των παραγόγων αυξάνει το συστημικό κίνδυνο δεν είναι σωστή. Τέλος, μήπως οι μικροεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να την χάνουν διαφορετικής μεταχείρισης. Αυτό εξαρτάται από το κατά πόσον πιστεύετε ότι μεγάλες εταιρείες δημιουργούν τον συστημικό κίνδυνο. Εάν η Επιτροπή σας δέχεται ότι ο συστημικός κίνδυνος δεν αφορά μόνο τις μεγάλες εταιρείες, τότε δεν τίθεται καν το ερώτημα. η Επιτροπή σας και το Συμβούλιο πρέπει να καταλάβουν ότι οι περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες δεν δημιουργούν συστημικό κίνδυνο, μεταξύ των οποίων και η χρήση των παραγόγων. Και η Επιτροπή Γεωργίας της Αμερικανικής Γερουσίας τα ίδια συμπεράσματα κατέληξε. Ελπίζω κι εσείς να καταλάβετε ότι οι ορισμοί που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να βασίζονται στην πραγματική οικονομία. Και αναμένω και η ΕΣΜΑ να μπορέσει να δικαιολογήσει την ύπαρξη εξαιρέσεων από τους κανόνες που θέλει να επιβάλλει. Ελπίζω να καταλάβατε ότι πρόκειται για προσπάθειες μείωσης του κινδύνου τα παράγωγα δηλαδή και όχι για αύξηση του συστημικού κινδύνου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχω συλλέξει τα ονόματα αυτών οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο και να θέσουν ερωτήματα. Θα ομαδοποιήσουμε λιγάκι τους ερωτώντες και ξεκινώ πρώτα με τον εισηγητή τον Βέρνερ Λάγκεν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες που μας έδωσαν μια πάρα πολύ επίκαιρη επισκόπηση της κατάστασης στα θέματα των εξοχρηματιστριακών παραγόγων και πέραν αυτών που ελέγχθησαν από τους εκπροσώπους του κλάδου, θέλω να πω ότι χωρίς να έχουν συγκρουστεί ανάμεσά τους, έχουν παρουσιάσει όλο το φάσμα της προβληματικής. Είναι σαφές και συμφώνησαν όλοι ότι χρειάζεται μια καλύτερη ε, ρύθμιση και κανείς δεν το αμφισβήτησε αυτό. Το θέμα είναι όμως ήδη τι μπορεί κανείς να τυποποιήσει. Να τυποποιήσει τα προϊόντα, τις διαδικασίες ή μονάχα το νομικό πλαίσιο. Θα πρέπει να επεξεργαστούμε το θέμα αυτό περισσότερο και η Κομισιόν βρίσκεται μονάχα στην αρχή της διαδικασίας παρουσίασης προτάσεων ιδίως για τους φορείς συμψηφισμού με κεντρικό αντισυμβαλόμενο. Πόσο μακριά πρέπει να πάει αυτή η τυποποίηση και μέχρι πού θα φτάσουμε με τις επιχειρήσεις, οι οποίες καλύπτονται συνήθως με διμερή συμψηφισμό. Το θέμα των κεντρικών φορέων συμψηφισμού επίσης ελέγχθη στην αρχή ότι είναι χρήσιμο σε κάθε περιοχή νομίσματος να υπάρχει τουλάχιστον ένας τέτοιος φορέας κεντρικού συμψηφισμού. Μετά όμως τίθεται το θέμα του αριθμού αυτών των, φορέων, το ποιο ακριβώς θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για αυτούς τους φορείς, το θέμα του ανταγωνισμού μεταξύ τους, το θέμα της διαλειτουργικότητας επίσης αναφέρθηκε, Μήπως η διαλειτουργικότητα οδηγεί και σε μεγαλύτερο κίνδυνο ή θα είναι καλύτερα να έχουμε ένα κεντρικό μονάχα φορέα συμψηφισμού. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε ένα φορέα ή πολλαπλούς φορείς στον ευρωπαϊκό χώρο και ένας από τους συναδέλφους επίσης έθεσε το θέμα αυτό, το ερώτημα το οποίο θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η άποψη των εμπειρογνωμόνων για το θέμα αυτό. Θα μπορούσε κανείς να δει τι γίνεται στους ε, φορείς συμψηφισμού όπως το κάνει κανείς στην τράπεζα, σε μια τράπεζα. Υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε το ίδιο επίπεδο ε, διαφάνειες αυτούς. Μήπως θα έπρεπε οι οργανισμοί κεντρικού συμψηφισμού να έχουν την ίδια άδεια όπως και μια τράπεζα για την λειτουργία τους μετά στο θέμα της διαφάνειας. Υπάρχει συμφωνία μεταξύ μας, αλλά ελέγχεται από διάφορους ομιλητές ότι η διαφάνεια στην αγορά είναι καλή, διαφάνεια για τις ρυθμιστικές και υποπτικές αρχές, αλλά και διαφάνεια για όλους τους ανταγωνιστές. Αλλά πού θα πρέπει να θέσουμε το όριο μεταξύ της προστασίας δεδομένων και της διαφάνειας και κυρίως να μην θίξουμε την αποτελεσματικότητα και τη ρευστότητα. Δεν ελέγχθησαν επίσης πάρα πολλά για ένα πολιτικό τμήμα της προβληματικής των ε, εξοχρηματιστιακών ε, προϊόντων για τον κίνδυνο, τον πιστοτικό κίνδυνο αντισυμβαλωμένου. Θα ήθελα λοιπόν να έχω περισσότερες παρατηρήσεις για το θέμα αυτό, πώς αντιμετωπίζει το πιστοτικό κίνδυνος αντισυμβαλωμένου. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε ασφάλεια κινδύνου αντισυμβαλωμένου σε περιπτώσεις παραγματικά όπως της Ελλάδος. Κατά την άποψη λοιπόν των εμπειρογνωμόνων, είναι απαραίτητο να ρυθμίσουμε χωριστά τον κίνδυνο αντισυμβαλωμένου. Δηλαδή πέραν από τους γενικούς κανόνες. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο ήθελα να τους θέσω. Νομίζω ότι θα συλλέξουμε πολλές ερωτήσεις γιατί μπορεί να επικαλύπτονται. Πηγαίνω τώρα στον ε, σκιώδη συγητή από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αποβάλω κάποιες ερωτήσεις τα γρήγορα. Πρώτα απ' όλα, ακούγοντας τον Ζαν Πιέρ Ζωή, αν δεν σφάλω σε κάποιο σημείο, αναφέρθηκε σε ένα κεντρικό φορέα συμψηφισμού για τις περιοχές με ομοιογενές νόμισμα. Τι σημαίνει αυτό σε σχέση με το ευρώ και την ευρωζώνη. Και θα ήθελα να ρωτήσω τους ε, συνομιλητές μας τι πιστεύουν για το governance. Πώς μπορεί να διαρθρωθεί η governance, η διακυβέρνηση ε, του κεντρικού φορέα συμψηφισμού. Τελευταίο ερώτημα. Ποια δυνατότητα υπάρχει να επεκταθούν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών συμπεριλαμβάνοντας στις προδιαγραφές αυτές που αφορούν τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών όλα τα παράγωγα που αποτελούν το διαπραγμάτευσης και τα παράγωγα των ρυθμιζόμενων αγορών και εκείνα τα παράγωγα εκτός των ρυθμιζόμενων αγορών. Ευχαριστώ. Και Swinburne. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λάγκεν που διοργανώσατε αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πολύ καλό που μπορέσαμε να ακούσουμε τόσους πολλούς ομιλητές, αγορητές που έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα. Όπως και σε κάθε άλλη ακρόαση ε, αναφέρθηκαν τελικοί τελική χρήση και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έγιναν δύο πλήρεις παρεμβάσεις και δεν θέλω να αφαιρθώ. Δεν μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτά που ειδηπόθηκαν. Με ενδιαφέρουν τα άλλα δύο θέματα που εφήγησαν η πρόταση για ενιαίο ευρωπαϊκό αποθετήριο και ίσως κάποιοι από τους εμπειρογνώμους μπορούν να διαφωτίσουν. Αν δεν ήταν ενιαίο αποθετήριο, πώς θα μπορούσαμε να, να έχουμε καλύτερη ενημέρωση για τα παγκόσμια προϊόντα, για να έχουμε και καλύτερη πρόσβαση γεωγραφικά στα στοιχεία. Αναφέρθηκε και μια άλλη έννοια, διαφοροποίησης, ρύθμισης βάση τύπου προϊόντος, ε, ε όγκου χρηστών και κατά πόσο ρυθμιστικοί φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούν να εφαρμόσουν ευέλικτο μοντέλο και πώς μπορεί κανείς να καλύψει τις μη χρηματοστικές εταιρείες όπως είναι οι ενεργειακές εταιρείες με άμεση ρύθμιση μέσω παρόχων χρηματοστικών εταιριών και αν χρησιμοποιηθεί ένα ευέλικτο μοντέλο ότι αυτή η περιπτώση πώς κανείς μπορεί να καλύψει στρατηγικές των hedge funds. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να γυρίσουμε σε ένα πρώτο γύρο απαντήσεων τώρα. Θέλω απλώς να σας υπενθυμίσω ότι πολλές φορές τα θέματα των φορέων κεντρικού συμπισφυμού κεντρικού αντισυλλεμβαλωμένου έχουν ε, εγερθεί και τα θέματα των μητρών συναλλαγών επίση. Τα έθιξε αυτά ο κύριος ε, Ζουέ, είπε την προσωπική του άποψη, όχι την άποψη τη ε, Σίζαρ. Ίσως όμως θα μπορούσε το πάνελ να μας πει ποιοι είναι οι κίνδυνοι που νομίζουν ότι ενέχονται λόγω του γεγονότος ότι οι κεντρικές τράπεζες είναι υπάροχοι ρευστότητα στους φορείς κεντρικού συμψηφισμού τη στιγμή που πολλές, πολλά παράγωγα καλύπτουν, μάλλον διασκελίζουν ζώνες ενιαίου νομίσματος και οι ανταλλαγές ε, συναλλαγματικών υποχρεώσεων είναι μια τέτοια περίπτωση τι γίνεται όταν έχουμε παραδείγματος χάρη βασικά προϊόντα όπως το πετρέλαιο τα οποία αποτιμούνται σε δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι όλος ο συντηρησμός πρέπει να γίνεται στις ΗΠΑ, κάτι το οποίο θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει από μια τέτοια προσέγγιση. Είναι κάπως εξόφθαλμο λοιπόν. Ποια είναι τα επιχειρήματα λοιπόν που λένε ότι πρέπει πράγματι οι φορείς κεντρικού συμψηφισμού να βρίσκονται μέσα στη ζώνη του αντίστοιχου νομίσματος και όχι να προσπαθήσουμε να έχουμε μια πρακτική λειτουργία ώστε να μειώσουμε τα προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να ανακύψουν μέσω της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας αυτών των φορέων συμψηφισμού. Θα ζητήσω λοιπόν τον κύριο Ζουέ να απαντήσει πρώτος γιατί νομίζω ότι βρίσκεται πίεση χρόνου ούτως ή άλλως. Θα προσπαθήσω να σεβαστώ τα όρια. τα όρια που θέσατε και το χρόνο σας. Μπορώ να σας διασφαλίσω ότι στις Ηνωμένε Πολιτείες πάντοτε θα υπάρχουν πεδία αντιστάθμισης. Είτε το θεωρείτε τέχνη αυτό είτε όχι. εφόσον υπάρχουν συμβόλαια που θα εκφράζονται σε ευρώ, εφόσον η ρευστότητα θα διασφαλίζεται από κεντρική τράπεζα για να αντιμετωπίσει τις χρεοκοπίες ή τις παύσεις πληρωμών. Ε, θα υπάρχουν άρα και περιθώρια θα προβλέπονται περιθώρια που διαθέτει η Κεντρική Τράπεζα και εφόσον θα χρειάζεται πάντα να υπάρχει κάποιος που επαληθεύει τι προβλέπουν οι οίκοι συμψηφισμού τότε οποιοδήποτε οίκος συμψηφισμού στη ζώνη ευρώ θα διαθέτει αυτά τα αντίστοιχα περιθώρια για λόγους προφανής και πολιτικούς και λόγους κυριαρχίας. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, θα κάνουν ό,τι θέλουν. Έχουν τα δικά τους εργαλεία, άλλο αυτό. Έχουν το δολάριο, έχουν ορισμένους οίκους συμψηφισμού και εργαλεία πρέπει και εμείς να έχουμε δικά μας, στη δική μας ζώνη, για να μην εξαρτώμαστε τόσο πολύ και να είμαστε καλύτερα οργανωμένοι. Αυτή είναι η προσωπική και πολιτική μου γνώμη. Εφόσον αναγκαζόμαστε να κάνουμε και πολιτική πολλές φορές. Δεύτερον, για... Δεύτερον, λέγω, νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρχει αρκετή ελαστικότητα αλλά ταυτόχρονα ισότητα. Γιατί γνωρίζω ότι πρέπει να είναι καλυμμένοι οι διάφοροι οργανισμοί, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και να λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς. Ξέρετε ότι υπάρχουν ειδικές αγορές η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, πρέπει να υπάρχει κάποια ελαστικότης και για το συμψηφισμό. Για να απαντήσω τώρα στις παρατηρήσεις του κυρίου Λάγκεν που είναι, ήταν σημαντικές, πράγματι πρέπει να δούμε τι σημαίνει τυποποίηση, το είπαν και οι άλλοι ομιλητές, των διαδικασιών μέχρι που θέλουμε να φτάσουμε, όπως και ο Κέσαρ πρέπει και εμείς να δούμε με ποιον τρόπο ακριβώς θα γίνει ο συνδυασμός και ο συμψηφισμός. Είναι σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Λάγκεν. Για να είμαι ειλικρινής πρέπει να σας απαντήσω ότι οι ίδιοι κίνδυνοι υπάρχουν και με τη μεγάλη συγκέντρωση όπως με το μεγάλο κατακαιρματισμό. Και αν θέλουμε μεγάλη συγκέντρωση πρέπει όλα να είναι ορισμένα στην τρίχα και εκεί μπορεί να αυξηθούν οι συστημικοί κίνδυνοι. Έπειτα, προσωπικά είπα ήδη και πριν ότι οι οίκοι συμψηφισμού μοιάζουν, θα μοιάζουν στη λειτουργία τους με πιστοτικά ιδρύματα. και χωρίς να μπω σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, νομίζω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τους τελικούς χρήστες. Όσοι εκφράστηκαν ως τελικοί χρήστες είπαν πράγματα που τα παρακολουθώ και εγώ με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς και η οργάνωση Κέσαρ. Αλλά δεν είναι η ίδια η κατάσταση των οίκων συμψηφισμού. Το είπε και ο κύριος Λάγκεν. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση. Δεν θα συμψηφιστούν τα πάντα και για όλους. Πρέπει να δούμε τι εμπεριέχει συστημικό κίνδυνο και τι όχι. Τέλος. για τα, τις βοήθειες που δίνουν κυρίαρχα, τις βοήθειες που δίνονται ως κύριο του κυριάρχου χρέους. Τα credit default swaps είναι ιδιαίτερα δύσκολο θέμα, αλλά πρέπει και αυτά να συμψηφίσονται για να μπορέσει ο ρυθμιστής να έχει τις απαραίτητες πληροφορίες και νομίζω κύριε Λάγκεν ότι αυτό μπορούν να το κάνουν οι ρυθμιστές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είναι πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσω να είσαστε πιο σύντομοι στο μέλλον, αλλά ο κύριος Ζουέ πρέπει να φύγει και δεν πρέπει να απαντήσουμε όλοι σε όλα τα ερωτήματα κατά ανάγκη. Ξέρω ότι η κυρία Μάστες θέλει να λάβει το λόγο Μάστες. Κύριε Πόλσον, θέλετε και εσείς να λάβετε το λόγο. Καλύτερα λοιπόν να ακολουθήσουμε την ίδια σειρά για να μην χαθούμε στο διάστημα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για το θέμα των ε, ανταλλαγών συναλλάγματος. Έχω απόψη γιατί εκπροσωπώ ένα οίκο συμψηφισμού που εργάζεται από την ε, Σουηδία, από τη Στοκχόλμη και κάνει συμψηφισμό σε έξι διαφορετικά συναλλάγματα. Δεν έχουμε σχέση με τις κεντρικές τράπεζες σε κάθε μία από αυτές τις έξι χώρες, αλλά τα καταφέρνουμε πολύ καλά με τη διαχείριση κινδύνου, η οποία εμπίπτει στις ε, διαδικασίες μας. Έχω δύο σημεία τα οποία θέλω να θίξω εδώ. Πράγματι, τα χρήματα των κεντρικών τραπεζών είναι καλύτερα την νέα ασφαλέστερα, αλλά δεν είναι απαραίτητο να έχει, δεν είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει καλά ένα οίκο συμψηφισμού. Οι κανόνες πρέπει να έχουν γενικό χαρακτήρα, να εξασφαλίσουν ότι οι απαραίτητες διαδικασίες και η απαραίτητη πρόσβαση θα υπάρχει, αλλά δεν προϋποθέτουν κατά ανάγκη σύνδεση με μια κεντρική τράπεζα για τους οίκους συμψηφισμού. Δεύτερο, για την ισότητα ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Για μένα είναι της υψής της σημασίας η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να αντιμετωπίσει όλε τις χώρες σε επίπεδο ισότητος και να έχει τη δυνατότητα κανείς να λειτουργεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με έδρα σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης. Επομένως, ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας ουσιαστικά θα πρέπει να εξασφαλίζεται εξίσου για όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Να, να συμπληρώσω για τα άλλα ερωτήματα αν θέλετε, δεν είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε εφόλου του επιστητού. Απλώς αυτές που θεωρείτε ότι σας αφορούν, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε το λόγο σε όλους, γιατί υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Θα έχουμε άλλες τρεις φορές τόσες ερωτήσεις στη συνέχεια. Εντάξει. Δύο σύντομε λοιπόν απαντήσεις ακόμα. Αν θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση των ε, οίκων κεντρικού συμψηφισμού όπως και των τραπεζών. Όχι. Τα CCP έχουν ένα ειδικό ρόλο στην αγορά και επομένως θα πρέπει να υπόκειται σε ρύθμιση ειδική για αυτούς τους οίκους. Πολλές από τις πτυχές αυτής της ρύθμισης θα είναι παρόμοιες ή οι ίδιες ταυτόσιμες με αυτές που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, αλλά υπάρχουν και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι απαραίτητο οι οίκοι κεντρικοί συμπληφισμού να αντιμετωπίζονται χωριστά. Δεύτερον, αν θα έχουμε ένα οίκο συμπληφισμού κεντρικού αντισυμβαλωμένου ή όχι στην Ευρώπη, εγώ πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο να έχουμε πολλούς τέτοιους οίκους σε διάφορα μέρη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μπλάιβ. Στο πρώτο ερώτημα επανέρχομαι για τον κατακαιρματισμό των διαφόρων συμβαλωμένων ε, και το θέμα της κυριαρχίας. Τα αποθετήρια, τα εμπορικά και κεντρικοί φορείς δεν είναι το ίδιο πράγμα απαραίτητα. Αυτά τα κεντρικά μητρώα είναι βασικοί φορείς που αργούν στην αγορά και είναι, ε, συνομιλούν με τους άλλους εμπορευόμενους. Εδώ μιλάμε για αποθετήρια που ε, είναι κάτι διαφορετικό, που είναι αποθετήρια πληροφοριών. Άρα θα μπορούσαμε να λύσουμε το θέμα, το πώς αντιμετωπίζουμε τον επιμερισμό των πληροφοριών ε, γεωγραφικά, με απλό τρόπο. Είχαμε παράδειγμα πρόσφατα του DTCC, αποθετηρίου που έκανε μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία θα διέθεταν πληροφορίες σε οποιοδήποτε ρυθμιστικό δίποτε ουδήποτε κράτους που ήθελε να γνωρίζει κάτι. Βασιζόταν, εγώ έμαθα, ήρθα σε επαφή με ρυθμιστικούς φορείς όλο τον κόσμο και θεωρούσαν ότι υπάρχει συμφωνία ότι η διαβίβαση των πληροφοριών των εμπορικών στα αποθετήρια ε, τα εμπορικά, ανεξάρτητα αν είχαν σερβερ εδώ στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική, που είχαν το σερβερ, τα αποθετήρια, ήταν κάτι με το οποίο συμφωνούσαν. Και είναι και εφικτό αυτό για τη συμμετοχή αγοράς. Και τα εμπορικά αποθετήρια μπορούν να γίνουν κάτι αντιληπτό. Αν αυτά όμως δίνουν τις πληροφορίες, τους ρυθμιστικούς φορείς που χρειάζονται τις πληροφορίες. Άρα είναι επιλύσιμο το πρόβλημα αυτό. Τώρα για τα κεντρικά συμβαλόμενα μέρη. Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα. Να αποφύγουμε τον υπερβολικό κατακαιρματισμό. Χρειαζόμαστε βελτίωση της αποδοτικότητας για να μειώσουμε τον κίνδυνο. Εν γέννη, στόχος είναι ελαχιστοποίηση των διαφόρων κεντρικών αντισυμβελαμμένων. Εγώ θα έλεγα ένα αντισυμβαλόμενο κατά κατηγορία στοιχείου ενεργητικού που έχει ειδικά του χαρακτηριστικά κινδύνου. Δεν είναι θέμα γεωγραφικό που γίνεται συναλλαγή ή ο φορέας που εκτελεί τη συναλλαγή αυτός που καθορίζει το χαρακτηριστικό του κινδύνου. Εγώ συστήνω ένθερμα παρόμοια ρύθμιση των κεντρικών αντισυμβελαμένων στον κόσμο και στενό συντονισμό, ελαχιστοποιώντας όμως κατά κατηγορία στοιχείων ενεργητικού να μην έχουμε πολλαπλούς κεντρικούς αντισυμβαλλομένους ε, στις διάφορες περιοχές, περιφέρειες. Ένα ερώτημα μου απευθύνθηκε συγκεκριμένα, γιατί αφορούσε την παρέμβασή μου, για την ευέλικτη το ΣΥΠΗΝ προσέγγιση σχετικά με τον καθορισμό ποσοτικών στόχων για συστημικούς, συστημικά σχετικούς φορείς η JP Morgan είναι συστημικά σχετικός φορέας και χρειάζεται χ της 100 κεντρικός συμψηφισμός των πιστώσεων. Είναι κάτι εφικτό και ευκταίο. Γιατί, ένα, αποφεύγουμε κίνδυνο του να καθορίσουμε τι είναι τυποποιημένο συμβόλαιο ή επιλέξιμη σύμβαση. Φεύγει το κίνητρο και από τους κεντρικούς αντισυμβαλωμένους και από τις συμμετέχοντες στην αγορά να κάνουν τις επιχειρήσεις τους πιο περίπλοκες για να αποφύγουν την απέτηση να περάσουν από κεντρικό συμψηφισμό. Εάν ένα ποσοστό της δραστηριότητάς μου πρέπει να συμψηφιστεί και μόνο, περιορίζεται ο συνολικός κίνδυνος που αντιπροσωπεύω για το σύστημα. Αυτό μπορεί να το διαχειριστεί ρυθμιστικός φορέας και εγώ αποφασίζω ποια προϊόντα θα συμψηφίσω ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους και κατά πόσο μπορούν να συμψηφιστούν. Και είπα πετύχω το στόχο. Γιατί πιστεύω λοιπόν ότι είναι εφικτό. Για το σημερινό κόσμο που δεν έχουμε ρύθμιση που δίνει συνεχώς την εξουσία στις ρυθμιστικές αρχές να το κάνουν αυτό, ad hoc ακολούθηση συνδυάζοντας το Federal Reserve τον είπα, το FSA και άλλους φορείς και ζητούμε από τους εμπορευόμενους ή τους πείθουμε να κάνουν ακριβώς αυτό. Ανελήφθησαν κάποιες υποχρεώσεις από την κοινότητα των dealers τα τελευταία χρόνια για αυξανόμενα ποσοστά των δραστηριοτήτων τους να ε, περνούν από συμφισμό κεντρικά. Ε, δυστυχώς ήρθε αργά λίγη πρόοδος. Όταν χτύπησε η χρηματοστική κρίση δεν είχε επιληθεί το πρόβλημα. Αυτή η πρακτική όμως υπάρχει και εφαρμόζεται σήμερα ανεξέλεγκτα. Εγώ δεν διατείνομαι ότι δεν χρειαζόμαστε τη ρύθμιση. Αντιθέτω, λέω ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο ρυθμι... η η ρύθμιση για να ενισχύσουμε αυτό το μηχανισμό και να συμμετέχουν όλοι. Είναι κάτι εφικτό και ένθερμα το συμβουλεύω. Δεν θέλουμε οτιδήποτε τυποποιημένο διότι η αγορά ε, κινείται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Καλώς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιος άλλος από το πάνελ θέλει να λάβει το λόγο τώρα για κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Κύριε Έλμπεκ. μια σύντομη παρέμβαση για το θέμα των ε, φορέων κεντρικού συμψηφισμού, αν θα πρέπει να είναι ένα κατά νόμισμα και δεν ξέρω αν θα δείτε όλα αυτά τα θέματα, αλλά υπάρχει το θέμα της διακυβέρνησης των φορέων αυτών, σε αυτό ήθελα να μιλήσω. Αν θέλετε να το αναφέρω αργότερα, ευχαρίστως μπορώ να επανέλθω αργότερα. Για τους τελικούς χρήστες, κάποιος θα ήθελε να πει κάτι, κ. Ρέμπαν. επανέρχομαι σε αυτό το ερώτημα το οποίο έθεσε η κυρία Σουίνμπερν. Πώς διαφοροποιούμε επί τη βάση του όγκου συναλλαγών. Νομίζω ότι αυτό το οποίο ρωτάτε είναι αν μπορεί να υπάρχει ένα ευέλικτο μοντέλο. Κατά την άποψή μου υπάρχουν δύο κομβικά θέματα. Ένα από τα οποία αφορά τους τελικούς χρήστες και το άλλο αφορά τους ρυθμιστές. Το πρώτο ερώτημα που είναι για τον τελικό χρήστη είναι αν χρησιμοποιείτε τα παράγωγα για να μειώσετε τον κίνδυνο και αν μπορείτε να το καταδείξετε αυτό. Οι περισσότεροι θα πούνε βεβαίω, μπορούμε να το τεκμηριώσουμε ότι αυτή είναι η πολιτική μα, να μειώσουμε τον κίνδυνο. Το δεύτερο ερώτημα, το οποίο ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να το απαντήσει ο ρυθμιστή, είναι αν υπάρχουν πραγματικά στοιχεία που να καταδεικνύουν το συστημικό κίνδυνο σε μη χρηματιστριακού τελικού χρήστε. Και νομίζω ότι εδώ είναι δύσκολο να καταδείξουμε ότι μη χρηματιστηριακοί χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν συστημικό κίνδυνο όπως χρηματοπιστωτικοί φορείς. Επομένως νομίζω ότι υπάρχει η βάση για εξαίρεση. Νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω ναι για το πρώτο ερώτημα, ότι δεν δηλαδή δημιουργούν συστημικό κίνδυνο και ότι χρησιμοποιούν μονάχα για αντιστάθμιση κινδύνου τα παράγωγα οι τελικοί αυτοί χρήστες. Εντάξει, θα γυρίσω τώρα στα μέλη του Κοινοβουλίου γιατί μπορεί να έχουν ε, κάποια θέματα για τη διακυβέρνηση τα οποία τους ενδιαφέρουν. Ήθελατε να επανέλθετε κύριε για το πρώτο θέμα, για τους ε, κεντρικούς φορείς στην ε, περιοχή του ευρώ. Νομίζω ότι η κυρία ότι Μπλάθ ήδη έθεσε αυτό το ερώτημα, ότι υπάρχουν πολλές συναλλαγές σε βασικά προϊόντα που εμπλέκουν πολλά πολλαπλά συναλλάγματα. Θα ήταν επικίνδυνο να υποχρεώσουμε να υπάρχει ένας τέτοιος φορέας για κάθε τέτοιο για κάθε περιοχή νομίσματος. Δεν θα θέλαμε οι Ιαπωνέζοι να πούνε ότι ό,τι είναι σε γέν θα πρέπει να ε, συμψηφίζεται στο Τόκιο και όλα αυτά. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια απάντηση σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας πω ποιος θέλει να λάβει τώρα ερωτήματα σε δύο ομάδες θα το κάνω για να μην είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Γιώκερ Κλούντ, Άννη Ποντιματά, Ούντο Μπούλμαν και η Κάθριν Στάιλερ. Αυτή θα είναι η πρώτη ομάδα. Και μετά Όλι Σμιτ, Πασκαλ Κέμπερ, Βίκυ Φόρτ και αν υπάρχει και κάποιος άλλος ο οποίος θες να θέσει ερωτήματα. Πασκάλ, είσαι σκιώδης συγητής. Ναι, δεν σας είχαμε ως σκιώδης συγητή. Θα σε βάλω στην πρώτη ομάδα τότε. Εντάξει. Ο κύριος Κλούτ. Σας ευχαριστώ και θέλω να ευχαριστήσω και τα μέλη του πάνελ για τις πληροφορίες που μας δώσανε. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Τονίσατε πάντα ότι υποστηρίζετε την διαφάνεια. Αλλά το έχετε σχετικοποιήσει αυτό λέγοντας ναι, διαφάνεια αλλά όχι υπερβολική διαφάνεια. Θα με ενδιέφερε να μου πείτε Πού είναι το πραγματικό όριο κατά την άποψή σας για τη διαφάνεια. Με ποιο τρόπο μπορείτε να το καθορίσετε αυτό πιο συγκεκριμένα. Είναι μονάχα ρητορικό σχήμα ή σημαίνει αυτό ότι θέλετε να διατηρήσετε το, το, το τωρινό status quo. Είμαστε συνηθισμένοι στους πολιτικούς οι οποίοι λένε καταρχήν συμφωνούμε, αλλά όταν ερχόμαστε στα συγκεκριμένα δεν συμφωνούμε. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πού θέλετε εσείς να θέσετε το όριο μεταξύ διαφάνειας και υπερβολικής διαφάνειας. Και το δεύτερο ερώτημα για τον εκπρόσωπο της E.ON. Εγώ κατανοώ την, τους κινδύνους που έχετε στην επιχείρησή σας που θέλετε να τους διαχειριστείτε και να τους μειώσετε. Και είπατε ότι και τα παράγωγα βέβαια έχουν χαρακτήρα ε, επικίνδυνο. Θα μπορούσατε να φανταστείτε κάποια εναλλακτική λύση για την αντιστάθμιση του κινδύνου. Να υπάρχει διαφορετική διαχείριση κινδύνου από ό,τι τη σημαίνει, η οποία δεν οδηγεί στο να γίνεται και αυτή η ίδια παράγον κινδύνου στις αγορές των παραγωγών. Ευχαριστώ. Εντάξει. Πασκάλ, αν θέλεις τώρα να λάβεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, ο Πασκάλ. Δύο ερωτήματα για τον κύριο Ζουγέ. Ιδιαίτερα για τον κύριο Ζουγέ. Το πρώτο ερώτημα αφορά το θέμα της διαλειτουργικότητας σε ποιο βαθμό, αν εμείς έχουμε, αν είχαμε ένα ή δύο μονάχα φορείς συμψηφισμού στην Ευρώπη, σε ποιο βαθμό θα πρέπει να είναι διαλειτουργικοί μεταξύ τους και με αυτούς που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν υπάρχει διαλειτουργικότητα με αυτές που είναι έξω από την Ευρώπη, κατά ποιε συνθήκες και με ποιο κίνδυνο. Και πώς θα αντιμετωπίσουμε το κόστος εποπτείας αυτών των φορέων, αν θα είναι διαλειτουργικοί. Δεύτερον, για τα credit default swaps. Είδαμε ότι στην πρόσφατη ιστορία, άμα πάρω το παράδειγμα της AIG, AIG μάλλον, της Αμερικανικής Ασφαλιστικής Εταιρείας, ο πολιτής ο οποίος είχε πουλήσει αυτά τα CDS τα οποία καλύπτανε την έκθεση, το άνοιγμα της AIG, δεν μπορούσε να καλύψει αυτές τις υποχρεώσεις ασφάλισης, δημιουργείται ένα συστημικός κίνδυνος. Επομένως υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αθέτησης για τα CDS και επομένως σαν ασφάλιση, σαν στοιχείο ασφάλισης τα CDS έδειξαν ότι είναι αναποτελεσματικά σε κάποιο βαθμό. Θα μπορούσαμε λοιπόν να φανταστούμε ότι όταν ένας χρηματοπιστωτικός φορέας εκδίδει CDS, είτε είναι ασφαλιστική εταιρεία είτε είναι τράπεζα, να υπόκειται σε κάποια δοκιμασία αντικσών συνθήκων, σε κάποια δοκιμασία αντοχής, που να δείχνει τι θα σήμαινε η αθέτηση του φορέα που παράγει τα CDS για το δικό του λογαριασμό και σε ό,τι αφορά την κάλυψη των κινδύνων που αναλαμβάνει μέσω των CDS. Γιατί αν δεν μπορεί να καλύψει αυτό τον κίνδυνο, δεν υπάρχει πραγματικά θεμητό δικαίωμα να πουλάει στην αγορά CDS. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψη των ε, μελών του πάνελ για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ιάννη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ζουγέ, στην ομιλία σας μιλώντας για την ε, κεντρική καταγραφή, για την ανάγκη κεντρικής ε, καταγραφής, χαρακτηρίσετε αφύσικο ε, το να μην μπορεί να έχει ο ρυθμιστής άμεση και άνεφόρων και προϋποθέσεων γνώση των πράξεων στις αγορές παραγόγων το, χαρακτηρίσατε μάλιστα ζήτημα ευρωπαϊκής κυριαρχίας και καθοριστικός ό,τι αφορά την αποτελεσματική διαχείριση των αγορών, σημειώνοντας ότι αυτό καταδείχθηκε ιδιαίτερα με αφορμή την κρίση του ελληνικού χρέους. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν και να ρωτήσω και τα υπόλοιπα αξιότιμα μέλη του πάνελ που έχουν διαφορετική άποψη. Ποιο ρόλο έπαιξε κατά τη, γνώση, κατά γνώμη σας η αγορά έξω χρηματιστηριακών παραγόγων και ειδικά των ε, CDS, Credit Default ε, Swaps, στην επιδίνωση της κατάστασης με το ε, ελληνικό χρέος και τι διαφορετικό θα μπορούσε να συμβαίνει σήμερα εάν είχαμε ήδη μια κεντρική υπηρεσία συμψηφισμού. Ευχαριστώ. Και τέλος, ο Ούντο Μπούλμαν. Κάθριν θα ξεκινήσει τον επόμενο γύρο. Ο Ούντο έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο συνάδελφος κύριος Λάγκε έκανε ένα αρχικό ερώτημα και το διατύπωσε ως εξή. Αν έχουμε συγκεκριμένους κανόνες τυποποίησης αναφορούν προϊόντα, διαδικασίες ή νομικό πλαίσιο. Ποιον από αυτούς τους μοχλούς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα. Εγώ δεν νομίζω ότι υπήρξε πλήρη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Θα ήθελα να επανέλθω στο ερώτημα αυτό και θα ήθελα να ξεκινήσω με τα προϊόντα, τα χρηματιστριακά προϊόντα. Υπάρχουν εκπρόσωποι του χρηματοοικονομικού κλάδου, τελικοί χρήστε, αλλά επίση υπάρχουν και αρμόδιοι για την εποπτεία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι, αν θέλετε, ο εκπρόσωπο των πολιτών ή των πελατών. Και το ερώτημα είναι τι νόημα έχει να πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με λογικό τρόπο τις τιμές των προϊόντων παραγματικά. Τι γίνεται όταν υπάρχει παραγματικά χάρη, όπως είπε ο αρμόδιος επότροπος, άνοδος της τιμής της βενζίνης επειδή υπάρχουν κερδοσκοπικές κινήσεις από πίσω και αυτό δεν έχει καμία σχέση με την προσφορά και τη ζήτηση. Το ίδιο γίνεται με τα αγροτικά προϊόντα. Υπάρχει μια διαφορά. Αν ανήκει κανείς σε ένα τομέα όπου παράγει τροφιμικά προϊόντα, και με τον τρόπο αυτό θέλει να καλυφθεί με τα παράγωγα ή αν κάποιο κάνει μια κερδοσκοπική δραστηριότητα σε βάρο των άλλων, οι οποίοι είναι στην πραγματική οικονομία. Όταν υπάρχει αθέτηση πιστοτικών συμβολέων, πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι εξασφαλίσεις για κάτι τέτοιο, τα CDS, καλύπτουν ένα πραγματικό κίνδυνο. Όταν κανείς έχει πάρει ένα CDS για μια υποχρέωση ασφάλισης που δεν εμπλέκει αυτό τον ίδιο, τι νόημα έχει αυτό το πράγμα. Επομένως, με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε προϊόντα με διαφοροποιημένο τρόπο σε σχέση με το αν έχουν μία χρησιμότητα στο σύνολο της αγοράς ή όχι και εάν είναι προϊόντα τα οποία εμπεριέχουν μία καταστροφική δύναμη την οποία εμείς δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Καλώς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα στραφώ ξανά προς τον κύριο Ζουγέ για να μπορέσει να μιλήσει πριν να αναχωρήσει και μετά θα στραφώ στα υπόλοιπα μέλη του πάνελ. Κύριε Ζουέ, έχετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω εν συντομία, λέει, αλλά είναι εκτός μικροφώνου και τον ακούμε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω εν συντομία. Να είστε ήσυχοι, κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο. Όσον αφορά το ερώτημα του κυρίου Κλουτ, οι επαγγελματίες που είναι εδώ έχουν την άποψή τους. Η διαφάνεια έναντι των ρυθμιστών πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δυνατή. Θέλουμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Αυτό που αληθεύει είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είπε και ο Σπόλσον, έχουμε ισορρόπηση μεταξύ ρευστότητας και διαφάνειας. Διότι έχετε τις τάξεις μεγέθους που μπορεί να είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς τα πράγματα χωρίς να επηρεάζει συστημικά την αγορά. Και πρέπει να έχετε γρήγορα ρευστότητα για κάποιους χρήστες, εμπορευόμενους κλπ. Πρέπει να το αναλύσουμε αυτό, αυτή την εξαίρεση, στον τομέα αυτό, γνωρίζοντας βέβαια και κατανοώντας αυτό που λένε οι επαγγελματίες, αλλά για τους ρυθμιστές η διαφάνεια πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δυνατή. Το επαναλαμβάνω. Για να απαντήσω στον Πασκάλ Κομφέ, υπάρχουν δύο στοιχεία όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα. Θα πρέπει να το δεχτούμε αυτό, αλλά μία αύξηση του κινδύνου, διότι συνδέουμε ε, κέντρα συμψηφισμού, αυτό συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους. Και μετά έχουμε και διαλειτουργικότητα, μεγαλύτερη διασύνδεση Όσο περισσότερε διασυνδέσει έχετε, αυξάνεται και το κίνδυνο διάδοση κινδύνων χωρί να τα έχει εγγύσει ότι θα είναι αντίστοιχη η πρόσβαση. Κάτι που υπογράμμισε η έκθεση του κυρίου Λάγκεν και το είπα και εγώ στην εισαγωγή μου και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Έχετε και τεχνικά σημαντικά προβλήματα, νομικά προβλήματα ελέγχου, διαχείρισης, αντιμετώπιση του κινδύνου όσον αφορά το stress test από την πλευρά μου. Είμαι υπέρ αναφέρθηκε στην έκθεση του κυρίου Λάγκεν είναι ένα από τα μαθήματα που αντλούμε από την κρίση και κάνουμε stress test όσον αφορά τους διάφορους εμπορευόμενους και τη δυνατότητα των κέντρων συμψηφισμού να ανεχθούν τους διάφορους αντισυμβαλόμενους. Και στο ερώτημα που έθεσε η Ελληνίδα φίλη μας, Γι' αυτό είμαι υπέρ, είμαστε υπέρ του Σέζαρ, εντό του Σέζαρ υπέρ ε, συμψηφισμού και μηχανισμού ε, καταχώρησης που γίνονται στην αγορά αυτά τον, αυτή των παραγωγών. Για να απαντήσω στο, ερώτημά σας, το λέω, έχετε σήμερα έρευνες που διεξάγονται, έχετε τους ρυθμιστές που κάθε ρυθμιστής ασχολείται με τα στοιχεία που αφορούν τους διάφορους φορείς, αλλά δεν έχετε σφαιρική εικόνα όσον αφορά την ελληνική κρίση. Είναι μία από τις δυσκολίες που υπογράμμιζα. Και το συνέστημά μου, το προσωπικό, και κάποιες έρευνες το εξετάζουν αυτό, ότι αυτό ποσοτικά, ποσοτικά επηρέασε σημαντικά, αλλά δεν υπήρχε ενίσχυση θεωρώ σαφές αυτό το πράγμα για τους λόγους που ανέφεραν οι τελευταίοι παρεβαίνοντας Είτε το θέλουμε, οι αγορές έχουν κάποια τάση ε, να πέφτουν για την κερδοσκοπία. Πράγματι, υπήρξε μάλλον ενίσχυση ανεξάρτητη από τον όγκο των συναλλαγών και υπήρξε η ενίσχυση της ελληνικής κρίσης ανεξάρτητα από την τελική κρίση. Αυτό δεν είναι απόκειται σε μένα. Πιστεύω ότι η δυσκολία θα είναι να δούμε τι είναι χρήσιμο για τους εμπορευομένους της αγοράς. Και ποια είναι τα προϊόντα που είναι ενδιαφέροντα σίγουρα για τα χρηματοστατικά ιδρύματα, για κάποιους επαγγελματίες, κάτι που δεν αντιστοιχεί πάντα όμως την ανάγκη καλύψεως των κινδύνων. Από αυτή την άποψη υπάρχει απόκληση μεταξύ του ρυθμιστού, μεταξύ διαφόρων αντιλήψεων και προσεγγίσεων και μεταξύ των επαγγελματιών. Περισσότερο στο χρηματοστατικό κόσμο από ότι στον κόσμο των επιχειρήσεων των μη χρηματοστατικών θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτή τη διάκριση και γι' αυτό γνωρίζοντας και εδώ συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν από διάφορους προσώπους των επαγγελματιών, γνωρίζοντας ότι δεν θα είναι όλα τυποποιήσιμα, η απάντηση στο ερώτημα που τίθεται είναι πώς μπορούμε να είμαστε στο δυνατόν φιλόδοξοι όσον αφορά την τυποποίηση για τους ρυθμιστές. Αυτό πρέπει να εξετάσουμε. Ευχαριστώ. Εντάξει. Είχαμε λοιπόν αρκετά ερωτήματα σε σχέση με τη διαλειτουργικότητα, που είναι ένα μεγάλο θέμα. Ίσως τα μέλη του πάνελ λοιπόν θα θέλουν να πούν κάτι για αυτό και ίσως επίσης θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν και τις πτυχές της διακυβέρνησης που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των κινδύνων. Νομίζω και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει δυνητικά σημασία για μας. Κύριε Πόλσεν, θέλετε να επανέλθετε λοιπόν. Ναι, λέει Πόλσεν. Σας ευχαριστώ για τη διαλειτουργικότητα. Υποστηρίζουμε τον ανταγωνισμό στα θέματα αυτά και η διαλειτουργικότητα είναι ένα σημαντικός τρόπος να εξασφαλίσουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ οίκων συμψηφισμού ώστε να δώσει η αγορά τις καλύτερες λύσεις. Αλλά αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν θέματα κινδύνου τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μεγάλη προσοχή οι φορείς κεντρικού συμψηφισμού θα πρέπει να μειώνουν τον κίνδυνο και δεν πρέπει να τους επιτραπεί να αυξάνουν τον κίνδυνο. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει σωστή στάθμιση του πώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Θέλετε να πείτε κάτι και για τα άλλα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν, δεν είσαστε υποχρεωμένους προφανώς να το κάνετε. Για τα CDS, για τις ανταλλαγές υποχρέωσης αθέτησης κτλ, για για το θέμα των CDS. Εμείς δεν είμαστε στη διαδικασία συμψηφισμού των CDS. Ίσως είμαστε ο μόνος οίκος ο οποίος δεν ασχολείται με τα θέματα αυτά. Αλλά δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Σε γενική βάση όμως δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξουν ειδικοί κανονισμοί για ειδικά προϊόντα όπως είναι τα CDS. Νομίζω ότι οι κανονισμοί οι οποίοι θα θεσπιστούν τώρα θα πρέπει να έχουν ένα γενικό χαρακτήρα για να καλύπτουν όλα τα παράγωγα. Σας ευχαριστώ η Blythe. Θέλετε να πείτε κάτι για το ερώτημα για τα CDS. Νομίζω ότι μία όπου όλοι συμφωνήσανε είναι για το θέμα της διαφάνειας. Εμείς επιμένουμε να υπάρχει 100% υποχρεωτική διαφάνεια σε μία βάση εφικτή τεχνολογικά, ώστε να έχουν τις πληροφορίες οι ρυθμιστές. Εάν υπάρχει κάτι τέτοιο, νομίζω ερωτήματα του αν η δραστηριότητα της αγοράς μπορεί να θυγεί ή αν μπορούν να υπάρξουν καταχρήσεις ή αν μπορούμε να, να υπάρξουν να στραφούν κάποιοι εναντίον του συμφέροντος ενός κυρίαρχου κράτους. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία μπορούν να τύχουν έρευνας με έναν τρόπο ο οποίος θα μπορούσε να μας οδηγήσει ακόμα σε μια λύση και όχι να οδηγηθούμε σε απαγόρευση προϊόντων τα οποία έχουν ακόμα πλέον για την αγορά αλλά χωρίς να έχουμε τέτοιου είδους διαφάνεια δεν νομίζω ότι μπορούμε να απαντήσουμε υποφελώς τα ερωτήματα αυτά. Επομένως, και εδώ πρέπει να ρωτήσουμε το ερώτημα πόσο διαφάνεια φτάνει και πώς είναι υπερβολική. Η διαφάνεια μετά τις συναλλαγές θα πρέπει να υπάρξει προσεκτική μέρημνα για το ποιες θα είναι και οι συνέπειες για τους συμμετέχοντες στην αγορά αν υποχρεώσετε λοιπόν οι συναλλαγές τους να γίνονται δημόσιες πολύ γρήγορα, αυτό θα οδηγήσει στην αγορά να πάρει αντισταθμιστικέ αντίστροφε θέσεις με αυτούς. Επομένως, θα πρέπει να δούμε κάθε πότε πρέπει να γίνεται αυτή η διαφάνεια, για ποια προϊόντα, ποιο. <laughs> δύο η ώρα το πρωί να τα δώσει κανεί αυτά τα στοιχεία είναι ίσω υπερβολικά. Δύο η ώρα το επόμενο απόγευμα ίσω είναι καλύτερα. Επομένω, προβλήματα όπω μέγεθο συναλλαγών, συνολικέ συναλλαγέ, ε, μπλοκ κτλ. Όλα αυτά πρέπει να τα εξετάσουμε προτού καταλήξουμε σε μια απόφαση, η οποία δεν μπορεί να είναι βεβαιασμένη απόφαση. Και το τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να δείξω είναι το θέμα τη διακυβέρνηση και τη διαλειτουργικότητα. Έκανε ένα σχόλιο προηγουμένω ότι η διαλειτουργικότητα είναι γενικά κάτι το επιθυμητό, αλλά μπορεί να έχει και κινδύνους. Αν φέρετε σε επαφή διαφορετικά προϊόντα ή προϊόντα από διαφορετικούς χώρους που δεν έχουν συνεκτικά μεταξύ τους πρότυπα κινδύνου, τότε οδηγείτε σε ένα, οδηγούμαστε σε ένα ανταγωνισμό προς το χαμηλότερο κοινό παρονομαστή, προς τα κάτω. Είναι απαραίτητο να υπάρχει προηγουμένως η ισοδυναμία και η ομοιομορφία των προϊόντων για να λειτουργήσει η διαλειτουργικότητα. Επομένω, η διαλειτουργικότητα έχει νόημα για μένα μονάχα αν είσαστε σίγουροι ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα πρότυπα κινδύνου για κάθε φορέα κεντρικού συμψηφισμού είναι επαρκέ. Επομένω, προ το παρόν, εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν πρόωρο να πούμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται, αλλά εν καιρό ενδεχομένω θα μπορούσε να είναι μια βιώσιμη οδό. Σήμερα δεν νομίζω θα ίσχυε κάτι τέτοιο. Τέλο, για τη διακυβέρνηση του κινδύνου. Εγώ πιστεύω ότι ένα από τα βασικά σημεία τα οποία τα ξεχνάμε πολλέ φορέ είναι ότι ο, κίνδυνος κίνδυνο αθέτηση από ένα κεντρικό αντισυμβαλόμενο θα πρέπει να βρίσκεται μέσα σε έλεγχο και σε όρια. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις όπου η βασική ιδέα είναι ότι αν υπάρξει αποτυχία, αθέτηση από τον κεντρικό αντισυμβαλόμενο, τα μέλη του ομίλου αυτού του φορέα συμψηφισμού θα πρέπει να έχουν ανοιχτή υποχρέωση να καλύψουν το, να καλύψουν το ποσό που δεν μπορεί να καλύψει ο κεντρικό φορέα. Ξαναγυρίζουμε όμω τότε στο μηδέν. Δηλαδή, φτιάχνουμε ένα κεντρικό φορέα για να κεντροποιήσει τον κίνδυνο που δεν, που δεν πρέπει να επιτρέπεται τι διαδικασίε. Ένα από του λόγου που εμεί θέλουμε να υπάρχει έλεγχο είναι ότι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτού του φορεί θα πρέπει να έχουν μια συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Αυτοί που χρησιμοποιούν λοιπόν του κεντρικού φορεί συμψηφισμού θα πρέπει να έχουν ένα ρόλο στη διακυβέρνησή του για να εμποδίσουν μηχανισμού οι οποίοι θα μπορούσαν να αποβούν σε βάρο του κοινού συμφέροντο ή των συμμετεχόντων στου φορεί κεντρικού συμψηφισμού. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να προσθέσετε εκεί κάτι, κύριε Ελμπάιτ. Νομίζω ότι η Μπλάθ το κάλυψε πολύ ωραία για το θέμα της διαλειτουργικότητας. Το μόνο πράγμα το οποίο θα σας έλεγα είναι ότι ο στόχος μας εδώ θα πρέπει να είναι ισχυρή, καλά ρυθμισμένη, φορείς κεντρικού συμψηφισμού. Ο ανταγωνισμός είναι καλός όταν είναι θετικός ανταγωνισμός και όχι αγώνας προς τα κάτω, ανταγωνισμός προς τα κάτω. Νομίζω ότι η διαλειτουργικότητα θα πρέπει να έχει το νόημα της συνεκτικότητας των υποδομών ώστε να μπορεί να υπάρχει καλύτερη ε, συνεργασία και ανταγωνισμός μεταξύ των φορέων κεντρικού συμψηφίσμου Αλλά προς το παρόν δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε πάντα προς την κατεύθυνση να υπάρχει κοινό ταμείο σε περίπτωση αποτυχίας και αθέτηση από τους, αόλους ε, τους κεντρικούς φορείς συμψηφισμού. Ναι. Θα ήθελα καταρχήν να σχολιάσω τη διαφάνεια και μέχρι πού πρέπει να φτάνει για μας θα έπρεπε να υπάρχει η ίδια διαφάνεια που υπάρχει με τα διάφορα επιμελητήρια για να μπορεί ο κόσμος να βλέπει σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει, ποιες είναι οι τιμές για ποιο προϊόν, αλλά δεν είμαστε και βέβαιοι. Βέβαια αυτές οι πληροφορίες πρέπει καταρχάς να δίνονται στους ρυθμιστές. Το συζητήσαμε με τη Γενική Διεύθυνση Ενεργείας και ειδικά καθεστώτα για την ενέργεια και για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος για να υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των αγορών. Όσο για τα αποθετήρια, νομίζουμε ότι τα αποθετήρια αναείδος δεν είναι κάτι που είναι ρεαλιστικό γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές και θα ήταν πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε εταιρεία να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους απαιτήσει. Θα ήταν όλα πολύ πιο εύκολα με ένα κεντρικό αποθετήριο. Τέλος, το ερώτημα του Ιαν, αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις στη χρήση των παραγόγων. Για μας εμείς θα θέλαμε μάλλον να υπάρχουν ρευστές και διαφανείς αγορές. Και το ίδιο νομίζω ζητάει η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Θεωρούμε ότι τα παράγωγα όμως είναι τμήμα της λειτουργίας μιας αγοράς. Άλλα εναλλακτικά προϊόντα δεν θα είχαν τόση διαφάνεια και θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για καινούργιες εταιρείες να μπουν στην αγορά. Νομίζουμε λοιπόν ότι τα παράγωγα είναι κάτι πολύ σημαντικό για την προστασία ακριβώς των καταναλωτών και καταναλωτριών. Θέλει κανείς άλλος να προσθέσει τίποτε, όχι λοιπόν. Α, ο κύριος Πόλσον θέλει να επανέλθει. Ναι, ένα σύντομο σχόλιο για το θέμα της governance. Κατ' εμέ, είναι πολύ σημαντικό τα κεντρικά και τα κεντρικά όργανα συμψηφισμού να είναι εκείνα που θα αντιδρούν σε, στη στιγμή που ξεσπάει κάποια κρίση. Αυτό βέβαια θα απαιτούσε ισχυρά και ανεξάρτητα όργανα. Πιστεύουμε ότι οι χρήστες δεν πιστεύουμε ότι οι χρήστες πρέπει να είναι τμήμα των διοικητικών επιτροπών. Ή μάλλον πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι και αυτοί τμήμα των διοικητικών επιτροπών γιατί δικά τους είναι τα χρήματα που χρησιμοποιούνται. Τελικά όμως πρέπει να είναι ανεξάρτητο, κυρίως ανεξάρτητο αυτό το κεντρικό σώμα συμψηφισμού. Συμφωνείς και εσύ. Ναι, να είναι ανεξάρτητα με εκπροσώπηση και των Χριστών, Αλλά και άλλων, όχι μόνο Χριστών. Μήπως θα μπορούσε κανείς να μας πει τίποτε πιο τολμηρό για τα credit default swaps διότι ορισμένοι συνάδελφοι είχαν κάνει ορισμένες δηλώσεις στον τύπο για τα credit default swaps ιδιαίτερα σε σχέση με το ελληνικό χρέος. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε αν θεωρείτε ότι το θέμα αυτό των credit default swaps δηλαδή έχει τύχει κάποιας κατάχρησης, είναι όλα γνωστά ή υπάρχουν και άγνωστα. Δεν μπορώ να σας προσθέσω πολλά στη γραπτή παρουσίαση που σας έδωσα. Νομίζω ότι πρέπει η πληροφόρηση να χορηγείται στους ρυθμιστές. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Και με συγχωρείτε αν δεν μπορώ να προσθέσω λεπτομέρειες. Ε, θα το... Θα στραφούμε τότε προς το Eurostat. Μήπως η Deutsche Bank μπορεί να μας πει τίποτα. Αυτό το ανέφερε η Blythe στην παρουσίασή της ότι τα παράγωγα δεν μιλούν έλλειμμα είναι βασικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην αγορά για τη χείριση του κινδύνου. Η AIG βοήθησε στο να γίνει παιδί της κρίσης. Και είναι άδικο αυτό. Είναι σκληρό να κατηγορούν τα προβλήματα για την προβλήματα της Ελλάδας στην αγορά των παραγόγων αυτών, των CDS. είναι το πώς αντιλαμβάνεται κανείς το θέμα, το πρόβλημα της Ελλάδας. Είναι λίγο σκληρό να παρουσιάζεται με διαφορετικό τρόπο το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Λυπούμε που σας στρίμωξα, γι' αυτό είμαι εδώ όμως. Προχωράμε και πάμε στον τελικό γύρο των ερωτήσεων. Μόνο την Κάθριν Στάιλερ και τη Βίκη Φόρντ έχω εδώ. Όλε και δεν είναι εδώ. Ο Σβέν επίσης θέλει να παρέμβει. Κάθριν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ το πάνελ των ε, ομιλητών. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των credit default swaps. Συζητήθηκε εκτενώς ο διαχωρισμός εκείνων που χρησιμοποιούνται για ασφάλιση, ο Ντο Μπούλμαν, ο κ. Λάγκερ και ο κ. Κανθίν αναφέρθηκαν σε αυτό, και εκείνων που χρησιμοποιούνται για κερδοσκοπία αποκλειστικά. Αυτά που χρησιμοποιούνται για ασφάλεια πρέπει να είναι κάτι καλό, αλλά αυτά που χρησιμοποιούνται για προφανή κερδοσκοπία είναι κακά και κανείς δεν αναφέρεται εδώ στο ελληνικό χρέος. Συμφωνείτε με αυτή την προοπτική ή διαφωνείτε. Άμεσο ερώτημα προς τον Blythe Masters. Την Blythe Masters. Περιγράφεσαι σαν η γυναίκα που κατασκεύασε όπλα μαζικής καταστροφής και, ανα... και δημιούργησε και διάφορα πιστοτικά παράγωγα. Και υπάρχει ένα κεφάλαιο του πώς έγινε κατάχρηση σε ένα βιβλίο, πώς έγινε κατάχρηση αυτών των μέσων. Βάσει των όσων γνωρίζεις τώρα, τι θα έκανες διαφορετικά παλιά. Καλώς. Εντάξει. Η Βίκη Φόρντα κολυφή. Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή που το οργάνωσε, οργάνωσε αυτή την ακρόαση μαζί με τη γραμματεία. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και ευχαριστώ και τους ομιλητές για το κόστος στον τελικό χρήστη. Γιατί ήρθαν ορισμένοι και μου είπαν ότι αυτό θα οδηγήσει το κόστος των ενεργειών αντιστάθμισης κινδύνου στα ύψη. Εγώ δεν καταλαβαίνω από πού βγάζουν τα αριθμητικά του στοιχεία. Γιατί είναι το κόστος του κεφαλαίου για τις τράπεζες ή κάποιες ε, υποθέσεις για το τι είδους εγγύησεις θα πρέπει να κινητοποιήσουν. Κανείς δεν μου έχει πει τι κεφάλαιο τι εγγυήσει απαιτούνται. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν έχετε κάνει κάποια ανάλυση σε βάση διαφόρων σενάριων για τις κεφαλαιουχικές απαιτήσει ή τις ανάγκες σε εγγυοδοσία που χρειάζονται για αυτή τη διαδικασία. Θεωρείτε ότι επίσης σε ό,τι αφορά τη Βασιλεία 2 οι συναλλαγές με τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους θα πρέπει να έχουν μηδενικό βάρος μηδενική στάθμιση κινδύνου. Πώς θα πείσουμε λοιπόν τον κόσμο να χρησιμοποιούν τους κεντρικούς αντισυμβαλωμένους και Μπλάθε εσύ είπες ότι αν μπορεί να υπάρξει μείωση κινδύνου σε διμερή συμψηφισμό που να είναι αντίστοιχη με αυτή των κεντρικών αντισυμβαλωμένων, θα πρέπει να υπάρχουν οι ίδιε απαιτήσει κεφαλαίου. Πώ μπορεί να καταλήξει λοιπόν στο ίδιο επίπεδο κινδύνου στο διμερή συμψηφισμό. Ευχαριστώ, δεν είσαι η τελευταία, γιατί ο Σβέλ, ο Σβέν είπε τελευταία στιγμή, θέλει και αυτός να ρωτήσει κάτι. Συγγνώμη, Βίκυ. Σε γενικές γραμμές έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξή: Πολλοί είπαν ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια εξαίρεση για τους τελικούς χρήστες. Προφανώς, έχοντας δει την πρόσφατη κρίση, υπήρξαν τελικοί χρήστες ή υποτιθέμενοι τελικοί χρήστες οι οποίοι ήταν κάπως εγκληματικοί στον τρόπο που συναλλασσόντουσαν. Αν δείτε την Ένρον, παραδείγματο χάρη, πώς συμπεριφέρθηκε. Επομένω το ερώτημα είναι μήπως πρέπει να υπάρχει κάποιο κατόφλι σε αυτό το χαρακτηρισμό των τελικών χρηστών και με ποιο τρόπο μπορεί να θεσπιστεί αυτό το κατόφλι ώστε να ξεχωρίσει τους πραγματικούς τελικούς χρήστες και τους τελικούς χρήστες που ουσιαστικά είναι τράπεζες επενδύσεων που συγχρόνως είναι και τελικοί χρήστε, Δεν ξέρω αν τα αγγλικά μου είναι αρκετά σαφή. Αλλά η Siemens, παραδείγματος χάρη, έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές στη Γερμανία σαν μια τράπεζα επενδύσεων που κάνει και κάτι ηλεκτρικά προϊόντα. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά στο παρελθόν είχε χαρακτηριστεί με αυτόν τον τρόπο. Το δεύτερο ερώτημά μου είναι τώρα κάπως πιο θεωρητικού χαρακτήρα. Άκουσα να λένε πολλοί από εσά όταν έλαβαν το λόγο ότι υπάρχει μια υποβόσκουσα υπόθεση ότι μεγαλύτερη ρευστότητα θα ευνοούσε την αγορά για να μπορεί να βρει τον καταλληλότερο τρόπο εγκατάστασης. Τουλάχιστον υπήρξαν πολλοί οι οποίοι επέκναν ορισμένε μορφέ ρύθμιση ω περιορίζουσε την ε, ρευστότητα. Το ερώτημα για μένα είναι το εξή. Από τη δική σα οπτική γωνία, υπάρχει κάποια ισχυρή επιχειρηματολογία ότι η μεγαλύτερη ρευστότητα οδηγεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τη αγορά. Εγώ μετά από πάρα πολλά από αυτά που είδα τα ακαδημαϊκά άρθρα για την ασυμμετρία πληροφόρησης και επίσης τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την έκθεση Turner, νομίζω ότι μπορεί κανείς να διαμφισβητήσει με πολύ καλά επιχειρήματα το αν είναι, αν απαραίτητα συσχετισμένη η μεγάλη ρευστότητα με την αποτελεσματικότητα της αγοράς. Βάσει της δικής σας εμπειρίας λοιπόν, θα ήθελα να ξέρω τι πιστεύετε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά από αυτά που ετέθησαν απευθυνόταν προς, τον Blythe, προς την Blythe Masters, οπότε στέχουν προς εσένα. Έχεις άλλο ερώτημα? Ε, συγητής έχει ένα ερωτηματάκι. Ένα κούτσικο ερώτημα για τις εξελίξεις των τελευταίων 10 ετών στα παράγωγα. Έχουν πολλαπλασιαστεί τα παράγωγα στην αγορά. Αυτό μπορεί να το δει κανείς από την πλευρά της, ε, του κινδύνου της αγοράς έχουν πολλαπλασιαστεί γιατί υποτίθεται ότι αυτό το απαιτεί η ανάγκη σε ρευστότητα της αγοράς. Θα ήθελα οι έξι εμπειρογνώμονές μας να πούν ποια είναι η άποψή τους σε σχέση με την πρόταση να υπάρξει μια αρρύθμιση η οποία υποχρεώνει την αγορά να επανέλθει στα επίπεδα του 2000 σε ό,τι αφορά τα παράγωγα. Γιατί έκτοτε έχουν αυξηθεί κατά κατά τέσσερις φορές τα παράγω από τρεις φορές το παγκόσμιο ΑΕΠ στο δωδεκαπλάσιο του παγκοσμίου ΑΕΠ. Είναι αυτό κάτι το οποίο είναι υπεύθυνο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να διατηρηθεί ή όχι. Καλώς. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πάει πίσω το ρολόι, πέντε λεπτά εκεί πάνω. Λοιπόν, Μπλάιδ, εσύ είσαι πρώτη. Ξεκινώντας λοιπόν με την φράση χρηματοπιστωτικά όπλα μαζικής καταστροφής. Αυτή τη φράση την ετοίμασε ένας περίφημος διάσημος επενδυτής, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός χρήστης παραγόγων ο ίδιος, ο Warren Buffett. Και βλέποντας το πλαίσιο που χρησιμοποίησε τη φράση αυτή και προσπαθώντας να καταλάβω πώς τα έβλεπε τα πράγματα, δοθήσεις της χρήσης των προϊόντων τους και της γνώσης που έχει, συμφώνησα με την άποψή του τελικά. Γιατί ε, με ποια έννοια. Πιστεύω ότι τα παράγωγα μπορούν να είναι πολύ επικίνδυνα και ενδεχομένω ε, πάρα πολύ επικίνδυνα μέσα αν τα χρησιμοποιεί ο λάθο χρήστη με, διαφορε... με λάθο τρόπο. Και ουσιαστικά αυτό ήθελε να πει, είναι σαν ένα σφυρί. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει με επικίνδυνο τρόπο ή με αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι και ένα χρηματοδοτικό μέσο. Αν δείτε τα αίτια των απολειών κατά την πρόσφατη χρηματοδοτική κρίση, είναι η δανειοδότηση παραδοσιακή, κυρίως ε, στα στεγαστικά δάνεια. Σε αυτό οφείλονται οι μεγαλύτερες απώλειες εν συγκρίση με τα παράγωγα. Παρ' όλα αυτά είναι θεμητό αυτό που αναφέρεται. Υπάρχουν μαθήματα που πρέπει να μάθουμε από την εμπειρία του ρόλου των παραγόγων κατά την χρηματοσυντική κρίση. Και όπως είπα και στην παρουσίασή μου, αυτά τα μαθήματα είναι σημαντικά να μαθευτούν. Και εγώ πρώτα απ' όλα Αισθάνομαι βέβαια ότι έμαθα από αυτή την εμπειρία και υπάρχουν κάποια πράγματα που θα ήθελα να τα είχα δει διαφορετικά. Όχι απαραίτητα να τα είχα κάνει εγώ διαφορετικά τα πράγματα, διότι ο ρόλος μου σε αυτό το τομέα είναι σχετικά πυρχιωμένος. Δεν θα προδώσω την ηλικία μου μπαίνοντα σε λεπτομέρειε. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά πυρχιωμένη η προσέγγιση. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν τρία-τέσσερα σημαντικά μαθήματα και πράγματα που θα ήθελα να δω να γίνονται διαφορετικά. Πρώτα απ' όλα, μιλώντας συγκεκριμένα για, το, ε, για την AIG, η AIG έγινε πολύ μεγάλος μέτοχος της αγοράς στον χώρο των παραγόγων. Ε, δεν ήταν ρυθμιζόμενος ο χώρος αυτός. Είχε συστημικές συνέπειες λόγω του μεγέθους και της κλίμακας των δραστηριοτήτων αυτή η εταιρεία, κυρίως στην πώληση της προστασίας πιστώσεων υπό τη μορφή παραγόγων πιστοτικών και κάποια ερωτήματα από τους ελέγχους διαχείρισης του κινδύνου και από τα στελέχη, τα ερωτήματα δεν ε, ε, τέθησαν ή δεν απαντήθηκαν επαρκώς. Ποτέ δεν θα πρέπει να θεωρηθούμε ότι μπορεί να γίνει ε, τόσο, μια τόσο μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κινηθεί χωρίς κάποια ρύθμιση και να, μην, να δημιουργηθούν συνέπειες που δεν εντοπίζονται. Αυτό είναι ένα μάθημα. Γιατί δεν παρατηρήθηκαν οι συνέπειες λόγω έλλειψης αναφοράς των παρα... παραγόγων, όχι μόνο CDS, αλλά σε όλα, τα στοιχεία του ενεργητικού. Η δραστηριότητά τους θα ήταν προφανώς ανησυχητική αν υπήρχε τρόπος ενημέρωσης και υποβολής αναφορών δεν θα συνέβαινε αυτό. Είναι το δεύτερο μάθημα. Υποχρεωτική ρυθμιστική υποβολή αναφορών και έλεγχος της κινήσεως των παραγόγων, να ξέρει ο κόσμος πού βρίσκονται οι κίνδυνοι, πού είναι οι συγκεντρώσει και πού βρίσκονται οι αρρύθμιστοι φορείς που αναλαμβάνουν υπερβολικούς κινδύνους. Τέλος, πέραν αυτού, υπήρχε μεγάλος βαθμός διασύνδεσης, όχι μόνο με την AIG, αλλά και με τους άλλους αντισυμβαλόμενους και μεταξύ αντισυμβαλωμένων της AIG. Και όταν έπληξε η κρίση, η ρευστότητα και η εμπιστοσύνη εξέλιπαν και ο ρυθμιστής υποχρεώθηκε να αναλάβει δράση παίρνοντας και χρήματα του φορολογουμένου, διότι φοβόταν τις συνέπειες και δεν ήξερε ποιες οι συνέπειες θα ήταν, εάν δεν λαμβάνονταν αυτά τα μέτρα. Αλλά αυτό είναι απαράδεκτο και γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ για να αποφύγουμε επανάληψη αυτού του φαινομένου στο μέλλον. Αυτό είναι το τελευταίο σημείο, δηλαδή το τελικό μάθημα που έμαθα. Δεν μπορούμε ποτέ να επιτρέψουμε τέτοιο βαθμό διασύνδεσης να είναι τόσο διαβρωτικός όπως κατά τη διάρκεια της χρηματοστικής κρίσης και όπως συζητήσαμε σήμερα. Πώς μπορούμε να το μειώσουμε αυτό αν αυξήσουμε σημαντικά το βαθμό στον οποίο ο κεντρικός ψηφισμός χρησιμοποιείται σαν εργαλείο στην αγορά παραγόγων για τη μείωση της διασυνδετικότητας. Αν όλα αυτά διορθωθούν, αν είχαν γίνει όλα αυτά δεν θα είχαμε το πρόβλημα της AIG και εκ βάθους καρδίας εύχομαι μακάρι να μην είχαν γίνει αυτά. Ένα άλλο ερώτημα ήταν τεχνικής φύσεως. Τι εννοούσα λέγοντας bilateral collateralization. Τι είπα, αν είπα κλήρη, έκανα λάθος. Διμερή παροχή εγγυήσεων ε, είναι ευρέως διαδεδομένη πρακτική, bilateral collateralization, στα παράγωγα όπου ε, δίνουν κάποια περιθώρια, κάποια ασφάλεια ε, οι διάφοροι αντισυμβαλόμενοι. Μπορεί να είναι υπομορφή ρευστού, κάτι που ε, μπορεί να γίνει και με ένα κεντρικό αντισυμβαλόμενο. Καμιά φορά όμω έχει τη μορφή περιπλοκοτέρων διευθετήσεων. Θα ήταν φυσιολογικό, παραδείγματο χάρη, μια τράπεζα που εμπορεύεται σε ενεργειακά προϊόντα με μεγάλη εταιρεία να κάνει καταγραφή των, ε, τα προϊόντα αυτά να τα πάρει σαν εγγύηση ή κάποιο εξοπλισμό σαν ε, εγγύηση και να διανοδοτεί βάση αυτού. Αυτά είναι κάποια τα εργαλεία που υποτίθεται χρησιμοποιούν οι τράπεζες για να δανειδοτούν την οικονομία, να τη βοηθούν να αναπτυχθεί, να παρέχουν ρευστό και μέσω αυτών των κανόνων περί κεφαλαίου δεν θα μπορεί ένας ε, να πάρει κανείς αεροπλάνο σαν εγγύηση κατά μιας, ε, έναντι μιας θέσεως σε, μια, ε, σε ένα χρηματιστήριο. Διότι δεν μπορεί να ρευστοποιηθεί ένα αεροσκάφο σε πέντε λεπτά. Γι' αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εγγύηση. Πολλοί προσπάθησαν να δεν τα κατάφεραν, τουλάχιστον επικερδός να ρευστοποιήσουν αεροπλάνο σε πέντε λεπτά. αυτό, ήταν, αυτό ήθελα να πω με το σχόλιο. Όμως όσον αφορά το θέμα τι γίνεται με εκείνους που παρουσιάζονται σαν τελικοί χρήστες αλλά είναι κακοί φορείς. Αυτό ήταν το ερώτημα, από ό,τι κατάλαβα, από το αξιότιμο μέλος περίπου εκεί. τι εννοούμε εκεί. Αν δημιουργούμε εξαίρεση για τελικό χρήστη, μήπως καταλήξουμε με κάποια κρυμμένα hedge funds ή μεγάλα χρηματοδοτικά ιδρύματα που αποκαλούνται τελικοί χρήστες και δεν είναι και κάνουν ε, πολλές συναλλαγές. Η απάντηση είναι ότι γι' αυτό χρειαζόμαστε υποχρεωτική αναφορά στους ρυθμιστές όλων των δραστηριοτήτων άνευ εξαιρέσεως και ρυθμιστή που έχει τη δύναμη να μπορεί να παρέμβει και να ζητήσει από τελικό χρήστη να δικαιολογήσει τη δραστηριότητά του και αν δεν ικανοποιηθεί τότε να αποσύρει την εξαίρεση. Αυτή είναι η λύση. Και κάποιο από του άλλου ομιλητέ ε, έκανε αυτή την ε, σύσταση με την οποία συμφωνώ απολύτω. Τέλο, όσον αφορά τη ρευστότητα και γιατί έχει σημασία και αν οδηγεί σε αποδοτικότητα, σίγουρα. Διάβασα πολλέ παρόμοιε μελέτε όπω και εσεί και υπάρχουν περιστάσει κατά τι οποίε τα δύο δεν ταιριάζουν. Εν γέννη, τα δύο ταιριάζουν. Παρόλα αυτά, αυτό που λέτε είναι σωστό. Δηλαδή, δεν είναι αποδοτική κάθε ρευστή αγορά. Όμω, καθοριστικό χαρακτηριστικό μια ρευστή αγορά είναι ότι μπορεί να πραγματοποιεί συναλλαγέ. Δηλαδή, μπορεί να μην συμφωνεί με την τιμή, αλλά υπάρχει μια τιμή που είναι εκτελέσιμη, διαθέσιμη, είτε αγοραστή είτε πολιτή. Και αυτή η έλλειψη ρευστότητα κλιμακώθηκε κυρίως κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστικής κρίσεως και οδήγησε στη διάλυση και στη δυσλειτουργία ε, του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος και υποχρέωσε τους ρυθμιστές ξανά να ακολουθήσουν την πορεία. Η ρευστότητα έχει σημασία διότι διατηρεί τη δυνατότητα του κόσμου να μπορεί να χειριστεί το κίνδυνο επομιζόμενος κινδύνους που τους αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια των φυσικών συναλλαγών ή που αναλαμβάνουν λόγω αποτυχίας κάποιου άλλου. Αν ένας μεγάλος, όπως η Lehman Brothers, ε, δεν τα πάει καλά, τι σημαίνει. Επομίζονται κάποιοι κινδύνους αγοράς που προστάτευσαν με την Λίμαν ε, που ήταν ε, συναλλασσόμενος. Και ο μεγαλύτερος κίνδυνος απέρευσε όχι διότι τους χρωστούσε χρήματα η Λίμαν και δεν πλήρωσε, αλλά η αδυναμία τους να βγούνε μετά από αυτή την θέση που είναι ένας κίνδυνος ε, αγοράς. Αυτά είναι τα σχόλιά μου. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ πλήρη αυτά που είπατε. Δεν ξέρω ποιος θα αντιμετωπίσει τώρα το θέμα του ζητήματος της μείωσης του όγκου και της συχνότητας ε, συναλλαγών στα, στα συμβόλαια παραγωγών. Mm. Ίσως ο συνάδελφός σας από την Deutsche Bank θα μπορούσε να πει κάτι τέτοιο. Με μεγάλη χαρά. <laughs> Ευχαριστώ, Μπλαϊφ. Για το θέμα αυτό που έχει να κάνει με τις αγορές. Μια αγορά που είναι υγιής είναι αυτή που υπάρχει μια υγιής ισορροπία μεταξύ αγοραστών και πολιτών. Εμείς δεν θέλουμε να αποκλείσουμε συμμετέχοντες από τις αγορές. Σίγουρα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει σωστή ρύθμιση για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά και ότι οι ρυθμιστές ξέρουν τι τους γίνεται. Είναι κάπως επικίνδυνο να αρχίσει κανείς να, αρχίζει, να σκέφτεται να αποκλείσει συμμετέχοντες στην αγορά όταν αυτοί έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν μέσα σε μια αγορά ο αριθμός τώρα των συναλλαγών στην αγορά των CDS υπήρξε τεράστια προσπάθεια να μειωθεί το ονομαστικό άνοιγμα το οποίο υπήρχε, το συνολικό άνοιγμα το οποίο υπήρχε. Το ονομαστικό, η ονομαστική αξία βέβαια αυτό το CDS είναι μια χρήσιμη έννοια αλλά δεν αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο. Είναι διαφορετικό ένα βραχυπρόθεσμο συμβόλαιο αθέτησης, ανταλλαγής αθέτησης με ένα αλφα ποσό ονομαστικό από ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο ανταλλαγής αφέτησης. Αλλά είναι χρήσιμο να υπάρξει αυτή η μείωση του ονομαστικού τη ονομαστική αξία σε άλλε κατηγορίε στοιχείων ενεργητικού, όμω όπω αυτή που εκπροσωπώ εγώ, θα πρέπει να γίνουν περισσότερε προσπάθειε να μειώσουμε το συνολικό ποσό. Εμεί έχουμε τα εργαλεία, απλώ θα πρέπει να το προσπαθήσουμε πιο δυναμικά. Μιλάμε λοιπόν για ονομαστική αξία. Ονομαστική αξία δεν είναι ο καταλληλότερος γνώμονας του κινδύνου. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερο να καταργήσουμε μερικά από τα συμβόλαια τα οποία συνάπτουμε. Ο κ. Ρέμπεν θέλει να λάβει το λόγο επίσης. Σε δύο σημεία, σε δύο ερωτήματα θέλω να επανέλθω που έφτιαξε η κυρία Φόρντ. Το κόστος για τους τελικούς χρήστες. Χωρίς αμφιβολία θα υπάρχει μεγαλύτερο κόστος για τον τελικό χρήστη που προκύπτει από το κόστος της χρήσης <clears throat> ρευστών στοιχείων εγγύησεως. Δεσμεύουμε λοιπόν χρήματα για να δώσουμε εγγύησει. αλλά επίσης και το κόστος για να διαπραγματευτεί κανείς νέους, ε, νέες διευκολύνσεις για αντιστάθμιση κινδύνου και τις δημιουργίες νέων τέτοιων φορέων. Θα χρειαστεί αυτό ώστε να δημιουργηθούν αυτοί οι φορείς. Ο μεγάλος, ο πραγματικός όμως κίνδυνος για μας είναι η διαδικασία της ε, Βασιλείας και η συζήτηση για τις, ε, για τις ε, απαιτήσει κεφαλαίου για τα παράγωγα και η, η αίτηση να, υπάρχει, να υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσει κεφαλαίου για μη κεντρικά συμψηφιζόμενα παράγωγα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι εάν οι Αμερικανοί δέχονται να υπάρχει ένα, μια εξαίρεση για τους τελικούς χρήστες. Αν το επιβάλλει η Ευρώπη αυτό θα είναι ένα πρόβλημα για μας. Αν η Ευρώπη εφαρμόσει τις, ε, τις ε, προτάσεις της Βασιλείας Όπω έχουν αυτή τη στιγμή, το πρόσθετο κόστο το οποίο θα πρέπει να απομισθούμε είναι πολύ μεγάλο και πάρα πολλοί τελικοί χρήστε θα πάψουν να χρησιμοποιούν εργαλεία αντιστάθμιση κινδύνου γιατί είναι τόσο μεγάλο το κόστο. Γι' αυτό εμεί έχουμε ζητήσει να υπάρξει μέσα στη διαδικασία διαβούλευση για την CRD4 και στην ε, διαδικασία τη Βασιλεία να τονίσουμε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί αυτή η πρόταση και να υπάρξει δυνατότητα να δοθούν εξαιρέσει για αυτού τους τελικούς χρήστες. Καταλαβαίνουμε ότι θα αυξηθεί το κόστος της διαχείρισης, αυτό είναι απαραίτητο για να ξεκαθαρίσει κάπως το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά αυτή η αύξηση του κόστου πρέπει να μείνει μέσα σε όρια. Θέλετε να λάβετε και εσείς το λόγο ή είχατε να πείτε κάτι, κάτι παραπάνω. Το μικρόφωνο παρακαλώ. Ένα σχόλιο για την περίπτωση ένρων που αναφέρθηκε προηγουμένως. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί με την ε, καλύτερη ρύθμιση για τα εξοχρηματιστηριακά παράγωγα. Εγκληματικές ενέργειες βέβαια δεν πρόκειται να αποφευθούν με υποχρεωτικό συμψηφισμό. Είχατε ζητήσει να λάβετε το... Ναι, <clears throat> ευχαριστώ. Για δύο ή τρία θέματα κύριε Πόλσον. Ξεκινώντας από αυτό που αναφέρατε προηγουμένως για το... την ισορροπία μεταξύ κινήσεων αντιστάθμισης κινδύνου εναντί της κερδοσκοπία πώς ξεχωρίζουμε τους καλούς από τους κακούς στον τομέα αυτό. Εγώ είπα ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο να το ελέγξει κανείς σε πρακτικούς όρους. Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος να αποφασίσουμε τι θα μπορούσε να είναι δυνητικά επικίνδυνο από συστημική άποψη εξαρτάται από το μέγεθος των φορέων. Είναι το μέγεθος το οποίο δημιουργεί κινδύνους και μπορείτε αυτό να το καταμετρήσετε με ποσοτικό τρόπο. Για το άλλο θέμα, για την στάθμιση κινδύνου των ε, φορέων κεντρικού συμψηφισμού μέσα στα πλαίσια της Βασιλείας σε ό,τι αφορά τις κεφαλαιοχικές απαιτήσεις. Παίζουν ένα σημαντικό ρόλο μείωση του κινδύνου αυτοί οι φορείς και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντική όταν θέλουμε να εστιάσουμε στη μείωση του κινδύνου. Νομίζω ότι η μηδενική στάθμιση για τα κεφάλαια αυτά θα είναι πραγματικά ένα έναυσμα, ένα κίνητρο για τους συμμετέχοντες στην αγορά να έχουν περισσότερο κεντρικό συμψηφισμό. Τέλος, κάτι ακόμα για το κόστος παροχής εγγυήσεων στους ε, φορείς συμψηφισμού. Ναι, αυτό προφανώς δεσμεύει χρήματα και η διαχείριση των κινδύνων από τους οίκους συμψηφισμού ζητά από όλους τους συμμετέχοντες να παρέχουν εγγυοδοσία και ενδεχομένω να την αυξάνουν όταν χρειάζεται αυτό. Αναρωτιέμαι όμω αν μπορεί κανεί να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο με άλλο τρόπο χωρί να υπάρχει κάποιο, κάποια εγγύηση για την προστασία μιας θέσης. Υπάρχει πάντα ένας, ένα κόστος. Το, ο κίνδυνος δεν μπορεί να δισταθμιστεί με μηδενικό κόστος χωρίς να υπάρχει κάποια εγκυοδοσία. Πιστεύω λοιπόν ότι οι οίκοι συμψηφισμού στην περίπτωση αυτή κάνουν την αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού πιο διάφανη και εξασφαλίζουν ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος με έναν τρόπο πειθαρχημένο. Είναι η ανάγκη να βγάλουμε τη μαύρη γάτα από την σκοτεινή αίθουσα και να τη δείξουμε σε αυτούς που είναι απ' έξω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζουέ. Ζητήσατε ξανά το λόγο. Πολύ σύντομα, για να απαντήσω διάφορες ερωτήσεις, λέει εκτός μικροφώνου ο κύριε Ζουέ. Είναι δύσκολο να κάνουμε διάκριση κάθε φορά τους τα καλά και κακά προϊόντα. δεν είναι να πούμε ότι το CD, τα CDS δημιούργησαν την ελληνική κρίση. Όμως είχαν στο ελληνικό έλλειμμα και ήδη ε, τα αξιόγραφα της ε, Ελλάδας είχαν ε, χρησιμοποιηθεί από διάφορους φορείς ήδη. Και ο ρυθμιστής πρέπει να φροντίσει για την αποφυγή της κερδοσκοπίας. Εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε σε αυτή τη φάση. Γι' αυτό είναι καλό ο ρυθμιστής να συνεργάζεται με τους εμπορευόμενους να κάνει κάποιες συστάσεις, να, κάνει, να υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης, καταγραφής και υποχρέωση συμψηφισμού και η, η περίπτωση σε AG είναι κάτι ξεκάθαρο. Εάν ανέχθηκαν αυτή τη μεγάλη ομάδα, ε, αυτό το μεγάλο όμιλο, ε, ε, σε αυτό οφείλεται. Θα έπρεπε αυτές οι επιχειρήσεις της αγοράς, ανεξάρτητο το μέγεθος, να πληρώνονται στη σωστή τιμή και ένα κόστο ετεπομίζονται οι χρηματοστικοί φορεί ανεξάρτητα τη δραστηριότητά του, αν είναι hedge funds, τράπεζα, οτιδήποτε άλλο και ο καθένα θα πρέπει να ασκεί τι δραστηριότητε του που τον χαρακτηρίζουν. Θα πρέπει να υπάρχει διάκριση δραστηριοτήτων χρηματοστικού τομέα. Ε, θα πρέπει να εξετάζεται τι γίνεται με τη φορολόγησή του και τι γίνεται με τι συναλλαγέ τη αγορά. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, όπω ε, το υπογράμμισε ένας από τους ε, παρεμβαίνοντες για τους χρήστες, τους τελικούς χρήστες. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε αντιστοίχηση της διατάξεων της Βασιλείας με τελικό κόστος. Στα πλαίσια της Βασιλείας ο ρυθμιστής το θέμα τι θα παρακινήσει με τους δικούς εμπορευμένους να πάνε προς τους 20 ψηφισμού. Μετά θα πρέπει να καθοριστούν τα όρια για τους τελικούς χρήστες, συναρτήσει τις εκθέσεώς τους και θα πρέπει αυτές οι εξαιρέσεις να αδειοδοτούνται όταν η έκθεσή τους δεν ξεπερνά ένα ορισμένο κατόφλιο το οποίο θα πρέπει να καθορίσουμε στα πλαίσια του Σέζαρ. Τρίτον, τρίτη πτυχή. Όσον αφορά τη ρευστότητα, συμφωνώ αρκετά με τα υποθέντα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αντιστοιχεία μεταξύ ρευστού και επίδοσης υποχρεωτικά τη οικονομική επίδοση ή τη ανάπτυξη απασχόληση. Αυτό παληθεύει από τη στιγμή όπου είμαστε σε μια κατάσταση όπου όλο και περισσότερο καταφεύγουμε στις αγο... καταφεύγουν οι μη χρηματοστικοί φορεί στην αγορά, θα πρέπει να προσέξουμε τη ρευστότητα των αγορών. Αυτό το αναγνωρίζω ότι υπάρχει θεωρητική συσχετισμό μεταξύ των δύο. Από τη στιγμή που υπάρχει αναταραχή μεταξύ τη χρηματοδότηση μέσω πιστώσεων εν συγκρίση των χρηματοδοτήσεων από την, συνάρτηση με τις χρηματοδοτήσεις από την αγορά πρέπει να προσέξουμε τι γίνεται με την τελευταία αυτής της αγοράς όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Τέλος, όσον αφορά τον όγκο των παραγόγων, αυτά που υπόθηκαν, ο κύριος Λάγκεν τα είπε όλα. Θα πρέπει να επανέλθουμε σε αναλογίες οι οποίες να είναι λογικές και με μηχανισμούς οι οποίοι φροντίζουν να έχετε σε αυτή, στις αγορές εκείνες που έχουν τριπλασιαστεί σε όγκο τις τελευταίες δεκαετίες για καλούς ή κακούς λόγους, θα πρέπει να επανέλθουμε στο ίδιο είδος οργάνωση όπως έχουμε και στις κανονικές χρηματοστητικές αγορές και στις αγορές των μετοχών. Και αυτό το σύστημα της διοργάνωσης θα πρέπει να είναι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζαμε στις αγορές των μετοχών σε σχέση με τις αγορές των παραγόγων που εξεράγησαν ε, και κατέρευσαν. Έχει και ο κύριος Λάγκεν, πρέπει να έρθουμε σε λογικά συστήματα πριν, που είχαμε πριν από την κρίση. Το βλέπουμε και από την επικαιρότητα της εβδομάδας. Διαφορετικά, αν κάνουμε κάτι άλλο, θα ε, καταλήξουμε σε διάφορα προβλήματα και κίνδυνο επαναλήψεως της ε, κρίσης. Αυτά λοιπόν έχω να πω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Τώρα για τα συμπεράσματα ο εισηγητής. Κύριος Λάγκεν. Θέλω εγώ να ευχαριστήσω και τους έξι ομιλητές του πάνελ. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων με πολύ μεγάλο βαθμό εμπειρογνωμοσύνης από τους ε, εισηγητές και αυτό νομίζω ότι έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία της νομοθετικής διαδικασίας στο Κοινοβούλιο. Έχουμε εμπλουτιστεί από αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα, Ακούσαμε τις έξι αυτές παρουσιάσεις και απαντήσεις από έξι διαφορετικά ε, από διαφορετικές οπτικές γωνίες και διαφορετικά πρίσματα, το συμπέρασμα που μπορούμε να βρούμε είναι ότι συμφωνούμε όλοι ότι απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια, ότι χρειάζεται να τροποποιηθεί ο τρόπος ρύθμισης σε όλα αυτά τα προϊόντα και ότι θέλουμε να έχουμε ανεξάρτητους οίκους κεντρικού συμψηφισμού αλλά σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες παραμένουν ακόμα πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία είναι αναπάντητα και κρεμή, Επομένως είναι δικό μας καθήκον μέσα στα πλαίσια της συζήτησης για τις εκθέσεις που εξετάζουμε τώρα η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων να διαλευκάνουμε αυτά τα σημεία και θα ήθελα να προτείνω στους ε, εμπειρογνώμονες να μας δώσουν και περαιτέρω τα φώτα τους σε ένα μεταγενέστερο επίπεδο και επίσης ευχαριστώ όλους για το γεγονός ότι καταφέραμε να τελειώσουμε εγκαίρως. Νομίζω ότι όλα τα ερωτήματα απαντήθηκαν, όχι πλήρως βέβαια, αλλά υπήρξε ένας μεγάλος αριθμός ερωτημάτων που απαντηθήκαν και θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές μας και τη γραμματεία και ελπίζω ότι από αυτή τη συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα έχουμε αντλήσει χρήσιμα συμπεράσματα από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εμείς προβλέπουμε στις 17 Μαΐου να ψηφίσουμε αυτήν την γνωμοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν και συμβασμοί οι οποίοι θα επιτευχθούν μεταξύ μα. Ο κύριο Μπαρνιέ είπε, ο επίτροπο Μπαρνιέ είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου θα παρουσιάσει η Κομισιόν τα πρώτα συγκεκριμένα μέτρα και μέχρι τότε θα πρέπει εμεί να έχουμε εγκρίνει αυτή τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ σε όλου λοιπόν. Um, Ωραία και εγώ σα ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν κάποιο θέλει να χειροκροτήσει το, πλάνε, το πάνελ. Άκουσα ένα να χειροκροτήσει, όσο μπορούμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Ωραία. Και τώρα εμεί θα προχωρήσουμε σε μια στην ανταλλαγή απόψεων για τις τροπολογίες της έκθεσης Langen. 17 Μαΐου δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι τότε θα προχωρήσουμε στο, στην ψηφοφορία. Θα πρέπει να ακούσουμε ποια είναι η επίσημη άποψη για τις ημερομηνίε, γιατί υπάρχουν συγκρούσεις με σημαντικά θέματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής για την κρίση. Θα μείνετε ή θα φύγετε. Θα, θα μείνετε. Α, ωραία. Ξαναδίνω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή σε αυτήν την περίπτωση. Θα συνεχίσω τότε, λέει ο εισηγητή, με πιο μπερδεμένα θέματα όπως είναι αυτό της αντιμετώπισης των τροπολογιών. Έχουμε το σχέδιο έκθεσης, το οποίο ήταν το σημείο αφετηρίας. Είναι σαφές ότι το αρχικό σχέδιο δεν μπορούσε να καλύψει όλα τα απαιτούμενα και γι' αυτό ευχαριστώ τους συναδέλφους οι οποίοι προσέφεραν μια σειρά από πρόσθετες προτάσεις και συστάσεις για την έκθεση αυτή. Θέλω να υπογραμμίσω καταρχήν ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ως Επιτροπή τροπολογίες διατυπωτικού χαρακτήρα. Τελικά, σε τελικό επίπεδο, θεωρώ δεδομένο, θα έχουμε σίγουρα στην έκθεση αυτή ένα διπλάσιο αριθμό συμπερασμάτων και διατυπώσεων από ότι στην τρέχουσα μορφή της έκθεσης. Αν δούμε τώρα τα λεπτομεριακά σημεία, εγώ, τα επιμέρους σημεία, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις τροπολογίες. Ένα και δύο παραπέμπουν σε προηγούμενα συμπεράσματα του Κοινοβουλίου και ομάδων εργασίας. Επίσης έχουμε στη συνέχεια μία σειρά από παραπομπές σε αιτιολογικές σκέψεις που αφορούν την ε, AIG, αλλά επίση τις ε, τιμές των βασικών προϊόντων, τα επιτόκια, το θέμα της χρησιμότητας των ε, παραγόγων κτλ. Ίσως εδώ θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική λύση που να καλύψει τις τροπολογίες 3 έως 6 και να φτάσει μέχρι την τροπολογία 9. Να κάνουμε λοιπόν μια αναδιατύπωση που να περιέχει όλες αυτές τις πτυχές που προαναφέραμε. Θα σας πρότεινα λοιπόν να κάνουμε κάτι τέτοιο και αυτή τη συμβαστική τροπολογία θα την επεξεργαστώ αυτή τη βδομάδα και θα την αποστείλω σε όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Μετά έχουμε το ένα δεύτερο σημείο που έχει να κάνει με την ιδιαιτερότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τροπολογία υπαριθμών 10, την οποία εγώ την καλωσορίζω, αλλά φυσικά αφήνει πολύ περιθώριο για αναδιατύπωση στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη μορφή. Τροπολογία 11, διεθνή πρότυπα. Απαιτεί, ζητά διεθνή πρότυπα αυτή η τροπολογία, τροπολογία 11, αλλά συγχρόνως θεωρεί ότι μπορούμε εμείς να προβούμε σε ευρωπαϊκά εγχειρήματα παράλληλα με τα διεθνή στάνταρ. Η τροπολογία 12 του κ. Γκοζές αναφέρεται στην στα στοιχεία που δίδει η Τράπεζα των Διεθνών Διακανονισμών στη Βασιλεία. Έχει αλλάξει κάποια στοιχεία λοιπόν και αν είναι πιο έγκαιρα τα στοιχεία του το, χαρακτηρί, το αποδέχομαι. Η τροπολογία 14 του κ. Κομφά αναφέρει νεότερες έρευνες σε σχέση με τα παραγωγά οι οποίες ζητούν να έχουμε πληροφορίες πιο αξιόπιστες για τα θέματα αυτά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε σε αυτή την έκθεση. Εγώ μάλλον Πιστεύω ότι θα πρέπει να απορρίψουμε αυτή την τροπολογία γιατί ξέρουμε ότι 15% των προβληματικών παραγωγών μονάχα είναι στις αγορές σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών. Έχουμε τη 15 του κ. Κλίντς, ο οποίος αναφέρεται στα θέματα της ανάπτυξης με το, με το θέμα της μόχλευσης και αυτήν την καλωσορίζω. Τροπολογία τώρα 16 Κράτσα, η οποία αναφέρεται στην ε, κερδοσκοπία με τα CDS που θεωρεί ότι είναι υπεύθυνη για το πρόβλημα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Ακούσαμε τώρα από τον κύριο Ζουέ ότι τα χρέη της Ελλάδος είναι πραγματικά και δεν οφείλονται στην κερδοσκοπία. κερδοσκοπία αφορά όχι μονάχα το, το χρέος αλλά και γενικά τη ζώνη του ευρώ. Από ό,τι γνωρίζω, ο όγκος των CDS για, τα για το ελληνικό χρέος ήταν περίπου το 1 τρίτο του συνολικού χρέους της Ελλάδος, όχι παραπάνω. Δηλαδή τα 2 τρίτα του ελληνικού χρέους δεν είχαν καλυφθεί από CDS. Επομένως δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να δημιουργήσει μια σχέση αιτία και αιτία του ότι τα CDS προκάλεσαν το ελληνικό χρέος. Περνάμε μετά στη θεματική της πολυπλοκότητος και της ανάγκης να καλύψουμε σωστά τον, κίνδυνο, τον πιστοτικό κίνδυνο αντισυμβαλωμένου. Εδώ υπάρχει γενική συμφωνία και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια δεύτερη συμβαστική τροπολογία η οποία θα συλλέξει όλες τις διατυπώσεις των συναδέλφων που θα καλύψει όλα αυτά τα οποία έχουν ζητήσει. Έχουμε μετά την τροπολογία 22 της Προέδρου μας, την οποία θα ήθελα να υποστηρίξω. Να υπάρξει έλλειψη διάκρισης στην πρόσβαση στα στοιχεία της, ε, των, ε, των αγορών και να υπάρξει σωστή λειτουργία των φορέων κεντρικού συμψηφισμού και εκεί ανακύπτει και πάλι το θέμα της ε, διαλειτουργικότητας. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο και ίσως πρέπει να το συζητήσουμε ακόμα περισσότερο πώς θα το διατυπώσουμε. Στη συνέχεια. Έχουμε προτάσεις πολλαπλές, ταυτόσιμες ουσιαστικά από διάφορους ε, συναδέλφους, οι οποίοι ζητούν το ίδιο πράγμα και μπορούν να αντιμετωπιστούν από κοινού. Θετικά όλες. Περνάω στην τροπολογία 26 της κυρίας Ποδηματά, η οποία αναφέρεται και αυτή στο θέμα της Ελλάδος και η διατύπωση όπως προτείνεται από την κυρία Ποδηματά στην ε, τροπολογία 26 νομίζω ότι μπορώ να την αποδεχθώ και πάλι δίνω μια θετική γνωμοδότηση για αυτή την τροπολογία. Το ίδιο ισχύει για την τροπολογία 28 του κυρίου Σκίνερ. 29 της κυρίας Μπάουλς τίθεται το ερώτημα του θα πρέπει να υπάρξει μια συστηματική αντιμετώπιση ή όχι. Ο κύριος ε, Κοζές έχει προτείνει στη συνέχεια μια διαγραφή παραγράφου. Είμαι κατά αυτής της ε, πρότασης και αντίθετα υποστηρίζω την τροπολογία της κυρίας Σουίνμπερν για την αντιμετώπιση ότι τα παράγωγα χρειάζονται λιγότερη ρύθμιση γιατί είναι θέματα που εμπλέκουν μονάχα τους εμπειρογνώμονες, αλλά αυτό φάνηκε και από τη σημερινή μας ε, ακρόαση ότι αντίθετα χρειάζεται πράγματι τα παράγωγα να την χάνουν μιας πλήρους ρύθμισης. Νομίζω ότι θα υπάρξουν πολλές τροπολογίες που θα συμπεριληφθούν στην τροπολογία συμβασμού υπαριθμών 3, τροπολογίες 29 έως 34. Στη συνέχεια, τροπολογία 35 έως 42. που αφορούν τους τελικούς χρήστες. Ένα θέμα που συζητήσαμε πλήρω σήμερα και που αφορά και τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι μπορούν όλες αυτές τις τροπολογίες να συνενωθούν σε μια συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 4. Έρχομαι στις τροπολογίες 37 του κυρίου Φέρμπερ, από τον οποίο θέλω κάποια ε, εξήγηση. Εγώ έχω βάλει ένα θετικό σήμα, αλλά δεν έχω καταλάβει τι λέει η τροπολογία του. Τροπολογία 40 στη συνέχεια. Τα στοιχεία, τα αριθμητικά, κατά την άποψή μου, είναι πολύ μικρά ότι τα μη χρηματιστιακά ιδρύματα καλύπτουν μόνο το 5 με 10% του συνολικού εμπορίου παραγόγων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της Κεντρικής Τράπεζας και της Κομισιόν είναι κοντύτερα στο 30% τα στοιχεία, το ποσοστό των μη χρηματιστιακών ιδρυμάτων, αλλά μπορούμε να το ξαναδούμε αυτό. Έχουμε τις τροπολογίες 43 έως 48 στη συνέχεια, οι οποίες και αυτές μπορούν να συγχωνευτούν σε μια συμβαστική τροπολογία και όπου μπορώ να δεχτώ την τροπολογία Swinburne, Όλι Smith και Swinburne, ενώ έχω προβλήματα με τη διατύπωση της κυρίας Γκουλάρ. Έχω προβλήματα. Αλλά, εν πάση θα υποβάλω μια συμβαστική τροπολογία. Στη συνέχεια, 49 και 50. Νομίζω ότι αυτές ζητούν την ε, διαγραφή του σημείου ε, αλλά υπάρχουν καλύτερες τροπολογίες άλλων συναδέλφων. Η τροπολογία 6 συμβαστική θα καλύψει την 51 μέχρι την 56 αφορά το θέμα των τελικών χρηστών πάλι και τα μη χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ότι χρειαζόμαστε περισσότερους κανόνες. Νομίζω ότι μπορώ να τις συνενώσω όλες σε μια συμβαστική τροπολογία και επομένως δεν χρειάζεται να υπάρξει ε, ούτε και μια χωριστή ε, ε, αξιολόγηση αυτών των τροπολογιών γιατί λένε περίπου το ίδιο όλες. Επίσης, στη συνέχεια έχουμε μια πλειάδα τροπολογιών 57, 58, 63, 64 65, οι οποίες μπορούν να μπουν στη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 7. Πρόκειται για τους οίκους ε, συμψηφισμού, ανταγωνιστικότητα, συστημική κίνδυνη και είναι εντυπωσιακό ότι και οι πέντε τροπολογίες αυτές προέρχονται από Γάλλους συναδέλφους. Από τέσσερις διαφορετικές πολιτικές ομάδες, αλλά <laughs> φαίνεται δεν υπάρχει μεγάλη σύμπνοια μεταξύ τους, αλλά παρόλα αυτά ελπίζω θα μπορέσει να υπάρξει κάποιο συμβιβασμός μεταξύ μας. Στη συνέχεια, περνάμε στις τροπολογίες. 67-68 και 59, οι οποίες από κοινού αντιμετωπίζουν παρόμοια θέματα, αφορούν την ε, ασφάλιση εναντί του πιστοτικού κινδύνου και την αντιμετώπιση τομέων όπως είναι ο ενεργειακός τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εφαρμογή αποφάσεων των G20. Ελπίζω και εδώ θα μπορέσει να βρεθεί μια διατύπωση, αλλά δεν έχει τελειώσει αυτό το εγχείρημα και έρχομαι στη συνέχεια στην τροπολογία 60 για την Ελλάδα, την οποία υποστηρίζω όπως την έχει διατυπώσει η κυρία Γκουλάρ. Γκουλάρ και όχι Γκουγιάρ. Δεν είναι Γκουγιάρ. Γκουλάρ. <laughs> Έχουμε στη συνέχεια τις προτάσεις του κυρίου Μπούλμαν και Ντομινίτσι. Μπορώ να τους δώσω θετική υποστήριξη. Είναι οι τροπολογίες 69, 62 και 61 και επίσης 59 εν μέρη. Ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό και πάλι έχουμε ταυτόσιμες γαλλικές και λίγο ιταλικές προτάσεις και έχω κάποιο πρόβλημα με την τροπολογία 73 κομφά η οποία, πώς να το πω τώρα αυτό, προβλέπει ένα πλαίσιο φορολόγησης αλλά πιστεύω ότι αυτό θα υπερεύαινε το, την εμβέλεια της ρύθμισης, γι' αυτό εγώ την, ε, εγώ την ε, απορρίπτω, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιος λόγος να το εξετάσουμε σε αυτή την έκθεση. 75 ε, μπέρες την υποστηρίζω, γιατί αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και ερχόμαστε στις τροπολογίες τώρα, 74 πάμε στις 75 με 83 που είναι πάλι γαλλικές και ταυτόσιμες και από άλλους έχουν κατατεθεί αυτές οι τροπολογίες που περιστρέφονται γύρω από το θέμα του σημείου 1 του εκτελεστικού τμήματος. Λένε ότι χαιρετίζουμε την πρόταση της Κομισιόν να υποβάλει τα εξοχρηματιστηριακά παράγωγα σε καλύτερη ρύθμιση με μητρώα συναλλαγών, με καλύτερη διαφάνεια κτλ. κτλ. Εδώ μπορούμε να τις συνδυάσουμε και να επελάβουμε τις διατυπώσεις όλων των συναδέλφων. Το ίδιο ισχύει για τις προτάσεις στο σημείο 1α που είναι οι 81-84, οι οποίες και αυτές είναι ταυτόσιμες με την εξαίρεση της 84 του κ. Όλη Σμιτ μπορούν να αντιμετωπιστούν με ενιαίο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και τις 87, θετικά τις υποστηρίζω όλες αυτές, 88 και έχουμε την 99 που αντιμετωπίζουν το δεύτερο, τη δεύτερη εκτελεστική παράγραφο να υπάρξει υποχρεωτικός συμψηφισμός των τυποποιημένων παραγόγων ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερος έλεγχος των κινδύνων. Εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις του Όλι Σμιτ, Τόμας Μαν, Γκοζές, Μπερές, Γκουλιά, Κουλάρ και όχι Γκουλιά, Δομινίτσι, Γκοζές, Σβίνμπορν, Κλίνς και Κονφέν και της κυρίας Μπόουλς. Όλες αυτές θα μπουν στην τροπολογία συμβασμού υπαριθμών 9. Τροπολογία 100 καράς. Ούτε και αυτή την κατάλαβα. Και εδώ ήθελα να, την, ε, να προτείνω την απόρριψή της αλλά δεν έχω μιλήσει ακόμα με τον κύριο Καρά. 101 κλίντς. Έχει όλες τις προϋποθέσεις για ένα συν, γιατί είναι σαφής και διαφανή αφορά το θέμα του λειτουργικού ελέγχου των εκτός χρηματιστηριών παραγωγών. 102 του κυρίου Καρά, δεν μπορώ να τη βρω τώρα που είναι ακριβώς. σημείο 3 του εκτελεστικού του που λέει ότι οι τιμές των παραγόγων θα πρέπει να αντανακλούν καλύτερα την ε, κατάσταση της αγοράς και το κόστος της υποδομής δεν πρέπει να καλύπτεται από τον φορολογούμενο αλλά από τους συμμετέχοντες στην αγορά. Και αυτό έχει κάποιο ιδεολογικό χαρακτήρα φυσικά. η πρότασή μου εδώ είναι να δεχτούμε την πρόταση αυτή του Τόμας ε, Μαν, της κυρίας Βίμπεν και του κυρίου Φέρβερ. Κλίντς και πάλι, ο οποίος θέλει να διαγράψει το σημείο 4 του ψηφίσματος, αυτό δεν το δέχομαι. Αντίθετα, η δέκατη συμβαστική τροπολογία καλύπτει τις τροπολογίες 108 έως 115, Μπάουλς, Κονφέν, Λάγκεν, πάλι Λάγκεν, Μπούλμαν, Δομινίτσι, Γκόζες, Όλι Σμιτ και Φαϊό, όλες μαζί. Πρόκειται για το θέμα του ότι πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ της ε, αντιστάθμισης κινδύνου στις επιχειρήσεις και της καθαρά κερδοσκοπικής δραστηριότητας χρηματαγορές. Αυτό ήταν σαφές και από την, ε, από την ακρόασή μας και η πρόταση της Κομισιόν λέει να υπάρξει διμερής συμψηφισμός αλλά με ιδιαίτερες απαιτήσει κεφαλαίου. Αυτό λοιπόν δεν ξέρω αν έχει νόημα να το ζητήσουμε από την Κομισιόν να αλλάξει. είδαμε ότι πολλοί θεωρούν ότι μια τέτοια ρήτρα μαζί με την εφαρμογή της Βασιλείας 2 θα είναι αντιπαραγωγική γιατί οι μη χρηματοοικονομικοί φορείς δεν επέχουν συστημικό κίνδυνο. Αυτό ήταν η τροπολογία συμβασμού υπορριθμού 10. Τώρα πάμε στην τροπολογία 116. Ντομινίτσι και Μπούλμαν την υποστηρίζω. Αφορά το συνολικό ε, όγκο των παραγωγών που θα πρέπει να μειωθούν μέσω μέτρων διαφάνειας και μέτρων για τον έλεγχο του κινδύνου αντισυμβαλωμένων. 1, 1, 7 και 118 των ιδίων αυτών κυρίων πάλι για μένα είναι στον ιδεολογικό χώρο ζητά να παρακολουθηθούν οι δράσεις ορισμένων επενδυτών σε σχέση με τα παράγωγα. Αλλά αυτό δεν είναι μια πρόταση που μπορεί να πάρει νομοθετικό χαρακτήρα ήδη την παρακολούθησε εγώ πρέπει να την απορρίψω. Είναι ψήφισμα αυτό, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε κάθε βλακεία σε αυτό το ψήφισμα. Έρχομαι στο σημείο 119 της κυρίας Γκουλάρ. Το είπα σωστά αυτή τη φορά. Για μένα πηγαίνει κάπως πολύ μακριά στο δεύτερο τμήμα. Αφορά την απόκτηση των καταλήλων πληροφοριών ώστε το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και η Εποπτική Αρχή για τις Αγορές να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ναι, εντάξει, το να, υπάρχουν, να υπάρχει διαφάνεια, ναι, αλλά όχι να υπάρξει εξονυχιστικός έλεγχος από αυτούς τους φορείς. 120 και 121, 122, 123, τέλος. Κλίντς, Καράς, Σφίνμπερν, Μπαούλς. Τις υποστηρίζω αυτές τις τροπολογίες. 124, Όλε Σμίτ, αφορούν το σημείο 6 και εδώ έχουμε τη συμβαστική τροπολογία 11 που καλύπτει όλους αυτούς τους κυρίους, Φίνμπερν, Γκοζές, Ντομινίτσι, Μπούλμαν κτλ. Και είναι ουσιαστικά μονάχα τροποποίησης διατύπωσης και εδώ θα πρότεινα μια συμβαστική τροπολογία η οποία θα απλοποιήσει τη διατύπωση. 130-131 Τις υποστηρίζω. Εδώ υπάρχει η υποχρέωση γνωστοποίησης από τους οίκους συμψηφισμού και τα Μητρώα. Και υπάρχει και το, πρό... το πρόβλημα που έθεσε η πρόεδρος, πώς θα αντιμετωπιστούν υποχρεώσεις προηγουμένων φορέων συμψηφισμού. Αλλά τονίζω και πάλι ότι δεν είναι εκεί το πρόβλημα αν το πρόβλημα είναι απλώ η προστασία εναντίον αντισυμβαλωμένων, γιατί πρέπει να καλύπτονται από του παλιού κανόνε για, την, για τον διψηφισμό. 1.3.2 3 1.3.7. Αυτή είναι η συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 12. Αυτό αφορά τι αρμοδιότητες τη ΕΣΜΑ, του Ευρωπαϊκού Εποπτικού Φορέα για το συμψηφισμό που έχει να κάνει και με τις τρίτες χώρες εδώ δεν ξέρω αν υπάρχει ήδη μια σωστή απόφαση. Νομίζω, απάντηση νομίζω ότι ο κύριος Μπάλτς για, τις, ε, για τους οίκους κεντρικού αντισυμβαλωμένου, συμπισφυρμού κεντρικού αντισυμβαλωμένου, να υπάρχει μια άδεια τράπεζας. Επομένως να υπόκειται στις ίδιες απαιτήσει κεφαλαίου όπως και οι τράπεζες. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα άξιζε να το συζητήσουμε και ο κύριος Μπάλτς δεν είναι παρόν. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να τεθούν στη συμβαστική τροπολογία 12. 1.38 για τα, τη χρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα, ναι. 139-140, δεν καταλαβαίνω πολύ καλά. Είναι η τροπολογία Βόρτμαν τροπολογίες Call και Μπάτς και μάλλον πρέπει να τις απορρίψω. Αφορά τις απαιτήσει ιδίου κεφαλαίου, αλλά αυτά είναι θέματα που αφορούν τον έλεγχο των τραπεζών και δεν νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούν εδώ. Αλλά ίσως μπορούμε να τις περιλάβουμε στη συμβαστική τροπολογία. Έρχεται η τροπολογία συμβασμού 13 για το σημείο 8, Bowles, Langen, Swinburne και εδώ έχω αναγκαστεί να αλλάξω εδώ την άποψή μου. Είχα γράψει το σχέδιο έκθεσης ότι η διαχείριση του κινδύνου, το σύστημα διαχείρισης κινδύνου, τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου δεν πρέπει να είναι σε ανταγωνισμό μεταξύ τους και δεν πρέπει να συμμετέχουν σε αυτά ή συμμετέχονται στην αγορά. Αυτό νομίζω πρέπει να το αναθεωρήσουμε. Τώρα λέω ότι δεν πρέπει να ελέγχονται πλήρως από τους ε, χρήστες τα οι και κεντρικού συμπλησμού, ούτε στι ΗΠΑ γίνεται αυτό. Επίσης θα πρέπει να παίζουν κάποιο ρόλο στην ε, ανάλυση κινδύνου αλλά αυτό να μην οδηγεί σε ανταγωνισμό προς τα κάτω. Αυτό τουλάχιστον κατάλαβα από αυτά που μας είπαν οι εμπειρογνώμονες σήμερα και αυτό θα καλύψει τις τροπολογίες μέχρι την 148, 149. Όλα αυτά τα οποία βρίσκονται στο σημείο 8 λοιπόν μπορώ να τα περιλάβω και αυτά είναι καλύτερα από τη δική μου τροπολογία, η οποία ήταν ίσω υπερβολικά περιοριστική. 150 της ε. Προέδρου. Για τεχνικά, τεχνικά πρότυπα για τον υπολογισμό των περιθωρίων, την οποία υποστηρίζω. 1 και 51, 151 αφορά την, την εποπτεία της ΕΣΜΑ για το αν θα πρέπει να καλύπτει όλους τους φέροντες κίνδυνο αυτό είναι ένα παλιό θέμα στο οποίο και εδώ άλλαξα την άποψή μου ενώπιον των νέων στοιχείων και εδώ απορρίπτω την τροπολογία του κυρίου, είχα βάλει μείον στην τροπολογία του Μινίτσι, αλλά μπορώ και αυτή να την περιλάβω στην 13. 152 σκήνερ θετικό, θετική γνώμη. Και ερχόμαστε τώρα στα θέματα που έχουν να κάνουν με το σημείο 9 εισαγωγή ενός Ευρωπαϊκού Μητρώου για όλες τις εκτός χρηματιστηρίου ε, συναλλαγές υπό την αιγίδα της ΕΣΜΑ ώστε να προωθηθεί η διαφάνεια. Και εδώ και πάλι υπάρχει μια σειρά από τροπολογίες για τέταρτη φορά από Γάλλους συναδέλφους τεσσάρων πολιτικών ομάδων κάποιος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά lobbying από τους γαλλικούς φορείς. Εντάξει, πρέπει να σας διασκεδάσω και λιγάκι. Ναι. και εδώ πρέπει να βρούμε μια συμβαστική λύση για, την, για να καλύψουμε αυτά που βρίσκονται στη συμβαστική τροπολογία 14. Ja, ist in Ordnung. Ist okay. Gut. Ωραία λέει ο Λάγκεν την τροπολογία 162-165 για το σημείο 9 και εδώ πιστεύω ότι τίθεται το θέμα ότι όταν έχουμε εμπόριο όταν δεν είναι δυνατόν να τα πρότυπα παράγωγα να τυχάνουν εμπορία σε, κεντρικά, σε κεντρικές αγορές θα πρέπει να πηγαίνουν υποχρεωτικά σε συμψηφισμό ε, κεντρικού συμβαλόμενου. Αυτή ήταν η απόψη του κ. Σκίνερ. Ακολουθούν τροπολογίες 166 με το θέμα των διεθνών προτύπων και το ερώτημα του κατά πόσο στην Ευρώπη θέλουμε να προωθήσουμε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων συμψηφισμού. Αυτό το ζήτησε ο κύριος Κλίντς και ακούσαμε σήμερα ότι αυτό επέχει ένα κίνδυνο και υπάρχει και η άποψη πολλών που λένε ότι δεν θα ήταν καλό αυτό να υπάρχει διαλειτουργικότητα γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε νέους κινδύνους των οποίων τη διάσταση δεν μπορούμε σήμερα ακόμα να αποτιμήσουμε. Έχω σκεπτικιστική στάση λοιπόν, τροπολογίες 171, 172, στο σημείο 11. Πρέπει να τις ελέγξω επιπλέον. Και δεν υπάρχουν άλλες τροπολογίες στο σημείο 11. Σημείο 12 υπάρχει ένας αριθμός τροπολογιών 181-182 συμβαστική τροπολογία 15 εκτός από την τροπολογία του συναδέλφου Κόμφα η οποία πηγαίνει πολύ μακριά Όλε αυτέ λοιπόν θα μπορέσουν να τι εσωματώσω εκτό από τον κύριο Κονφέν. Κύριε Κονφέν, γενικά σε έχω ικανοποιήσει, αλλά δεν μπορώ να τα δεχτώ όλα. Πάμε στο 12α και το 12β. Υπέρ τη ε, τροπολογία Ντομινίτσι και Μπούλμαν. Έχω κάνει κάποιε μικρέ αλλαγέ. Θα βάλω θετικό πρόσημο σε αυτέ τι τροπολογίε. Συμβαστική τροπολογία 16 για την 184 μέχρι 190 στο σημείο 13. Υπάρχουν ευθυγραμμισμένες εδώ τροπολογίες που αφορούν θέματα που είναι λιγάκι διατυπωτικά. 191 όλοι Σμιέτ υπέρ για τον περιορισμό ε, παραγωγών που επέχουν συστημικό κίνδυνο, το ίδιο ισχύει για την 192, 193 του κ. Κομφέν, θετική γνωμοδότηση από τον εισηγητή, 194 Σφίνμπερν και ερχόμαστε στην 195 μέχρι 200 οι οποίες αφορούν το σημείο 14 και εδώ ασμένος θα δεχόμουν να παραμείνει το αρχικό κείμενο. Και θα, θα χώμα για αυτό το λόγο οι τροπολογίες. Έχω την 199 της κυρίας Μπερές, η οποία όμως μπορεί να γίνει δεκτή ως προσθήκη στο σημείο 14. Και το ίδιο ισχύει και για την 200. Όλοι Σμιτ. 17 Συμβαστή τροπολογία 201 έως 207 που αφορούν το σημείο 15 του ψηφίσματος και αφορούν τον, την ασφάλεια έναντι κινδύνων με ΣΕΔΕΕΣ. Έχουμε λοιπόν τροπολογίες από 7 συναδέλφους οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν και να συνενωθούν. Και στη συνέχεια ερχόμαστε στην τροπολογία 208. Άλλο ερώτημα τίθεται εδώ. Αμάν. Συγκέντρωση αγοράς. 80% των παραγωγών CDS εκδίδονται από 6 μεγάλες εταιρείες. Αυτά είναι τα στοιχεία δεσμένα. Δύο από αυτά τα έξι ιδρύματα ήταν παρόντα σήμερα. Η JP Morgan, που είναι το μεγαλύτερο και η Deutsche Bank που είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εκδότης. Υπάρχουν άλλες εταιρείες όπως η Morgan Stanley και η Goldman Sachs. Και το ερώτημα είναι αν πρέπει να κάνουμε κάτι για να αντιμετωπίσουμε την υπερσυγκέντρωση της αγοράς. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η πρόταση δεν είναι πρέπουσα και επομένως την τροπολογία αυτή της κυρίας Μακάρτη την απορρίπτω. 209 μπερές θέλει η κυρία Μπερές την ευρωπαϊκή διάσταση να την έχει σε επίπεδο CCP φορέων και δικού συμψηφισμού. Αυτό λέει και η τροπολογία 211 Μπούλμαν και Ντομινίτσι. Και τώρα 210 της κυρίας Μπάους η οποία λέει ότι τα ΣΕΝΤΕΣ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, σε μια χώρα νομίμως ακόμα και αν δεν έχουν εκδοθεί από κρατικές αρχές. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τώρα δεν είναι απαγορευμένη η χρήση αυτών των CDS, αλλά όταν πρόκειται για κρατικό χρέος στη ζώνη του, του ευρώ, ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο για τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν για τα κατόφλια επί τη βάση των οποίων πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Αυτά είναι θέματα ε, επίμαχα που δεν τα έχουμε ακόμα συζητήσει. Επίσης, Ντομινίτσι και Μπούλμαν λένε ότι θα πρέπει να περιορίζονται τα CDS σε ένα όγκο δανείων και μόνο. Δηλαδή να μην ξεπερνούν την έκθεση σε δάνεια. Στη συνέχεια. Έχουμε τις τροπολογίες για το short selling, για την γυμνή πώληση, για την επιβολή ορίων και τις ε, δημόσιες δραστηριότητες σε σχέση με την εμπορία στα χρηματιστήρια. Ντομινίτσι, δεν ξέρω αν μπορούμε να λύσουμε τα θέματα αυτά σε ναι, σχέση ναι. με τις τοπικές πωλήσει, αλλά για τα ανώτερα όρια έχουμε τις τοπολογίες Bowles, Langen και Dominici. Είμαι υπέρ αυτών. Αλλά για τον κύριο Κομφέν με σπαραγμό καρδιάς δεν μπορώ να την υποστηρίξω την τροπολογία του 216 γιατί ζητά η Κομισιόν να προβεί σε μια ανάλυση κόστου ωφέλου σε σχέση με τη χρηστοσυντία στα τελευταία δέκα χρόνια, όταν έχει δείξει η χρηματοοικονομική κρίση ότι δεν είναι πολύ αποτελεσματικά κτλ. Και ότι δεν είναι αποδοτική λοιπόν η αγορά. το σταθερή. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν νομίζω ότι αυτό είναι δίκαιο και θέλω να απορρίψω. Να θεωρήσω αυτό το σημείο ως απερχαιωμένο. 218 Ούλμαν Ντομενίτσι. Για τη 218 λοιπόν, τι να σας πω, τι θα καλύπτεται σύμφωνα με τη ρύθμιση όλα τα παράγωγα υψηλού κινδύνου, συμφωνούμε, αυτή είναι η διατύπωση, ότι θα καλύπτονται αυτά, όλα τα παράγωγα και τα παράγωγα των εταιριών. Αυτό είναι κάτι που αξιολογείται διαφορετικά στις διάφορες τροπολογίες που υποβάλλονται. 18 συμβιβαστική 18 από τη 18 και μετά έχουμε προτάσεις Ντομινίτσι, Μπούλμαν, Όντε Σμιτ, Γκοζές, Κλίντ, Ποδηματά, Γκοζές, Ντομινίτσι, Ιμπερές και Μπούλμαν. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά πιστεύω ότι μπορούν να ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι τροπολογίες. Διάκριση μεταξύ χρηματοπιστωτικών και μη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μπορούμε να καταλήξουμε σε λογικό συμβιβασμό, συμβαστική 18, για τη συμβαστική 18. Στο τέλος έχουμε διάφορες ε, συστάσεις να συμπεριλάβουμε την παράγραφο 17 και να επεκταθεί μάλιστα 17, να συμπεριληφθούν και άλλα προϊόντα. Έχουμε καλές συστάσεις της κυρίας Γκουλάγα και του κυρίου Γκοζές, του κυρίου Μπούλμαν και της κυρίας Μπερέ. Αναφέρεται εδώ, αναφέρεται λέγω εδώ, η διακοπή της έβριθης λειτουργίας. Εν γέννη εγώ είμαι ανοιχτός για οποιαδήποτε πρόταση σχετικά με το θέμα. Οπότε πλησιάζουμε στο τέλος. Έχουμε και κάποια άλλα σημεία. Έχουμε και άλλα σημεία, λοιπόν, που πρέπει να καθορίσουμε, να βάλω και συν στη 2.26, τροπολογία 2.26, Βέρμπερ, 2.36 μαλλον βερμπερ Φέρμπερ, 17α, 17β. Έχουμε κάποιες τροπολογίες και εδώ. Παρόμοιες είναι, παρεμφερείς. 17α, θετική άποψη, 18 θετικό πρόσημο, να ενθαρρύνουμε συντονισμό σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά χρειαζόμαστε και το ευρωπαϊκό επίπεδο και ρύθμιση και σε αυτό. Πρόταση Bowles, Dominici, Bullman, Gouges και Κομφά. 2.49 φτάσαμε στη 2.49 της κυρίας Γκουλά που καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι ευρωπαϊκοί και μη ευρωπαϊκοί ρυθμιστές να έχουν πρόσβαση στα αποθεματικά, στα κέντρα απόθεσης και ε, στα κέντρα ε, καθάρισης ε, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμοιβαία πρόσβαση στην, στις πληροφορίες, κέντρα συμπληφισμού μάλλον εντός, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τα παράγωγα, υπάρχει μια ρύθμιση στη ΣΥΠΑ για ε, τα κέντρα συμψηφισμού και αν δώσουμε πρόσβαση στους Αμερικανούς θέλουμε και εμείς πρόσβαση στα δικά τους κέντρα συμψηφισμού. Καλωσορίζω λοιπόν αυτή την πρόταση. Λογική πρόταση. Και τέλος μια τροπολογία της κυρίας Γκουλάγ που υπογραμμίζει τη σημασία τακτικής αναθεώρησης της αποτελεσματικότητας των μελλοντικών ρυθμίσεων με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην αγορά και να γίνεται ιδέως προσαρμογή όποτε είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Είμαι υπέρ μιας τέτοιας εμπόριο σε αγροτικά προϊόντα και σε, άλλο, σε άλλα προϊόντα. Έχουμε προτάσεις σχετικά πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε μια σωστή προσέγγιση ειδικά με αυτό και να διευθετήσουμε το θέμα. Εγώ ανέφερα μόνο συγκεκριμένα κάποιες τροπολογίες. Μόνο κάποιες τροπολογίες ανέφερα. Θα προσπαθήσουμε, θα προσπαθήσουμε λέγω να λάβουμε υπόψη αιτήματα των συναδέλφων, ανησυχίες αυτών και προσπαθήσουμε να προβληματιστούμε δεόντως εντό συμβαστικών προτάσεων. Και θα συντάξουμε το κατάλληλο κείμενο κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα και θα σα αποστείλουμε το κατάλληλο κείμενο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα όλα αυτά που μας είπατε βοήθησαν πολύ τους σκιώδεις εξών και εμένα. Δεν έχω εδώ τον κατάλογο των σκιωδών, αλλά μήπως ο κύριος Δομινίκη θέλει να πάρει το λόγο. Θέλει, όχι, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Θα περιμείνουμε να υποβληθούν οι συμβιβαστικές και μετά θα συζητήσουμε τότε εις βάθος με τον κύριο Λάγκεν. Καλά, τότε θα λάβω εγώ το λόγο. Είπατε ότι δεν είστε σίγουρος για μερικές από τις ντροπολογίες μου. Η 131 αφορούσε την εξαίρεση που είπατε και εγώ εννοώ ότι όταν κάτι έχει επιληθεί πριν γίνει κάνωση ψηφισμός πρόκειται για σχεδόν ταυτόχρονη λειτουργία και Κατανοώ ότι στη διατύπωση μπορεί να μην είναι σαφές. 186 Νότς. αναφέρεται στις απαιτήσει για κεφαλαια, κεφαλαιουχικές εγγυήσεις στη CRD 4. Η ΔΕ 210 προσπαθώ να πω ότι υπάρχουν και θεμητές χρήσεις των credit default swaps. Γι' αυτό είπα σημειώνει. Δεν προσπαθώ να πω ότι δεν μπορώ τίποτε άλλο. Μπορείτε να το ξανασκεφτείτε λοιπόν. Αν μια εταιρεία ενδιαφέρεται πολύ για να οργανώσει διακοπάς στην Ελλάδα, μπορεί τότε να θελήσει για να μην εκτεθεί πολύ, να χρησιμοποιήσει ένα credit default swap. Η 237. Εκεί Λέω ότι με τις 337 ε, λέω για τις άδειες εκπομπών μερικοί με ρώτησαν τι εννοούν όλα αυτά. Μα είναι θέμα που αφορά μάλλον την Επιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά είναι πολύ σχετικό και εδώ ως Επιτροπή Εικόν. Γιατί έτσι όταν μειώνεται κάτι ε, σφίγγει και η αγορά. Λοιπόν, αυτά ήταν οι δικέ μου. Σβένο Σκιώδη, θέλει να πει κάτι. Δεν είσαι Σκιώδη, είσαι ποιο είναι τότε. Α, ο Πασχάλης, εντάξει. Α, ο Πασχάλης, καλά. Φαίνεται κάτι έκανε λάθος πάλι η γραμματεία, τέλος πάντων, Πασχάλη. Όχι, ήθελα απλώ να τονίσω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις που είναι παρόμοιες οι γαλλικές τροπολογίες ενώ προέρχονται από διαφορετικές ομάδες, ε, δεν ισχύει αυτό για τις δικές μου. Άρα να μην μιλάει για όλες τις πολιτικές ομάδες που έχουν συνεννοηθεί ο κύριος Λάγκεν. Εγώ έχω την ίδια θέση με τον κύριο Ντομινιτσί να περιμένουμε τους συμβιβασμούς για να συζητήσουμε. Πούμε γιατί δεν μπορέσαμε όμως ακόμη να τα πούμε με τον εισηγητή. Και Α, ο κύριος Λάγκεν. Δεν πρέπει να σκεφτούμε μονάχα το θέμα των χρονοδιαγραμμάτων. Χρειαζόμαστε και 14 μέρες για να μεταφραστούν όλα αυτά. Και δεν νομίζω ότι εγώ σταμάτησα για, τα, για τις διακοπές του Πάσχα για να... και σταμάτησα την εργασία. Συγγνώμη. Όχι προς Θεού, προς Θεού. Όλοι έχουμε μεγάλο φόρτο. Ξέρω τι τεράστια εργασία ήταν αυτή η εξέταση των τροπολογιών, αναμένω και εγώ τους συμβιβασμούς. Με βάση όμως αυτά που είπαμε σήμερα αναρωτιέμαι μήπως ένα από τα θέματα δεν πρέπει να διαχωριστεί δηλαδή. Μπορεί να χρειαστεί στόχευση αναείδος επένδυσης. Αφού η αγορά των CDS έχει φτάσει το 95% πια. να ζητήσουμε από την Κομισιόν να το συμπεριλάβει. Μάλιστα, ο κύριος Φάρμπερ. Ευχαριστώ πολύ. Μου ζήτησαν να μιλήσω για την τροπολογία 37 παρόλο παρόλο που πρέπει να πω ότι συμφωνώ με τον εισηγητή έχει Έχουμε βάλει ένα συν και ένα πλήν, διότι έχουμε μία αντίθεση εδώ. Υπό το φως των όσων ακούσαμε όμως και προς τα εκεί που κατευθυνόμαστε, χρειαζόμαστε διαφορετικούς κανόνες ανάλογα με την περίπτωση. Γίνονται ανάλογα με το είδος του εμπορίου που γίνεται. Εγώ θα ήθελα να μας υποχρεώνουν να δικαιολογούμε βέβαια τις ε, τροπολογίες και θα ήθελα πολύ σε αυτή τη δικαιολόγηση των τροπολογιών ε, αυτή τη δικαιολόγηση να τη βρίσκουμε στο φάκελο. Διαφορετικά δεν καταλαβαίνω σε τι χρησιμεύουν οι τροπολογίες. Εγώ δεν... Έτσι νομίζω. Ούτε εγώ ούτε συνεργάτες μου βέβαια θέλουμε να ε, ετοιμάζουμε αιτιολογίες αν δεν τις βρίσκουμε να συμπεριλαμβάνεται. Εδώ τι λέμε, τι είναι τράπεζα, τι δεν είναι τράπεζα, ε, εγώ πήρα τον ορισμό του MIFID γιατί είναι ο ευφιέστερος ορισμός διότι δεν είναι στο... Ε, η τράπεζα δεν μπαίνει στους κανόνες του MIFID και αντίστροφα. Ο κύριος Λάγκεν σαν εισηγητής θα έπρεπε να υιοθετήσει αυτή την ε, τροπολογία κατά την άποψή μου. Ναι, μία εξήγηση να κάνω λέει ο κύριος Λάγκεν. Όχι, όχι, θα επανέλθετε σε λίγο. Όχι, όχι, πρόκειται περί τεχνικού προβλήματος κυρία Πρόεδρε λέει ο κύριος Λάγκεν. Στις, αιτιολογικές, στις ε, αιτήσεις πρωτοβουλίας δεν υπάρχουν πια αιτιολογικές εκθέσεις, μόνο οι νομοθετικές εκθέσεις έχουν ε, μια αιτιολογική έκθεση. Δεν προβλέπετε λοιπόν να έχουμε αιτιολογική έκθεση, αυτό ήθελα να πω. Thank Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τιμή στον κύριο Λάγκεν. Υπήρξατε εξαιρετικά πολύ άσχολος. Κάνατε διακοπές στο Πάσχα. Κάνετε διακοπέ για Πάσχα. Α, τότε κάτσε πολύ το Πάσχα. Όλα καλύπτονται. Η τροπολογία 200. Τι είπατε. Είναι ουσιαστικό αυτό. Θέλετε κατά περίπτωση να απαγορεύετε. Να απαγορεύονται κάποια μέσα. Α, αστιάκια, αστιάκια. Ναι, χρειαζόμαστε κάποια άλλη αστεία. Αν ακούσατε, ακούσατε κάποιες από τις επικρίσεις που ακούστηκαν στην ακρόαση, είσαστε υπέρ της απαγόρευσης. Εγώ θέλω να εξαιρεθεί αυτή η λέξη, να μείνει εκτός αυτή η λέξη. Ο κύριος Ουέ απάντησε. Είπε ότι δεν θεωρούσε ότι θα ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο και ξέροντας τι είπε εκείνος και τι είπε η γαλλική κυβέρνηση και λέγει, είναι στο πλευρό σας, κύριε Λάγκεν. Δεν μπορείτε να τους ακούσετε και σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι επικοδομητικό εργαλείο, γιατί 200 μιλάνε, ναι, γιατί 200. Είπε ότι ήταν υπέρ του ευρωπαϊκού, υπέρ της 200. Υπέρ αυτού του, της προτάσεως, λέει η Πρόεδρος. Είναι απλούστατο. Θέλετε απαγόρευση νέου. Ναι, Εγώ βλέπω να υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ της απαγόρευσης των CDS. Ο κύριος ε, Όλη Σμιτ θέλει κάτω από ορισμένε συνθήκε να υπάρχει μία προειδοποίηση και σε άλλε περιπτώσει απαγόρευση. Εγώ νομίζω ότι είναι αντιφατικέ αυτέ οι δύο αντιμετωπίσει. Για όλα αυτά τα οποία έχουμε αποφασίσει, προφανώ χρειαζόμαστε μία ε, πλειοψηφία. Είναι τόσο απλό, αγαπητέ συνάδελφοι. Όλοι Σμιτ. Όλε Σμιτ ήταν ο τελευταίο ομιλητή. Κανεί δεν μου γνέφει. Κύριε Λάγκεν, Τελειώσαν οι ομιλητέ, Αν θέλετε να ολοκληρώσετε τη συζήτηση με οδήποτε τυχόν σχόλιο. Θαυμάσια, σας ευχαριστώ όλους και ελπίζω ότι θα μπορέσει να κλείσει αμέσως τη συνεδρία πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Όπω Όπως μου λέγουν, διαπραγματευόμαστε την τελική ε, ημερομηνία για την ψηφοφορία. Οπότε πέρα στη συνεδριά σας. Έχουμε συνεδρίαση συντονιστών στις 18.30. και 30. σας βράδυ.